Morgen. Ich darf die unterbrochene Sitzung eröffnen und darf Sie herzlich begrüßen und willkommen heißen zur Fortsetzung der Sitzung des Haushalts. Καλημέρα σας. Άρχεται η σημερινή συνεδρίαση. Να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Προχωρούμε με την ημερήσια διάταξη με το σημείο 9, την ειδική έκθεση μέσω της αλλαγής 2011 για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας που παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιστημιστική ασφάλεια στην υποσαχάρια Αφρική. Εισηγητής ο Μπαρτ Στάς. Ο κύριος Βέσπεργκ είναι ο επί της ουσίας από το ηλεκτρικό συνέδριο. Να τον καλωσορίσω και θα ήθελα να του δώσω τον λόγο ως πρώτο μιλητή. Funktioniert es nicht, die Technik mit dem Mikrofon? Doch. sorry, I'm sorry for... Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι ενώπιόν σας. Θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση των κυρίων ευρημάτων και συστάσεων του ελέγχου απόδοσης για την αποδοτικότητα Τη αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιστημιστική ασφάλεια στην υποσαχαρή Αφρική. Λίγα λόγια για την ίδια την επιστημιστική ασφάλεια. Η επιστημιστική ασφάλεια ήταν και παραμένει ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Υπολογίζεται ότι ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι υποφέρουν από πείνα. Έχει οριστεί αυτό ως μια κατάσταση όπου όλοι και πάντοτε δεν έχουν αρκετή πρόσβαση σε αρκετή τι τροφή για μια ενεργό και υγιή ζωή. Η επιστημιστική ασφάλεια είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην υποσοχάρια Αφρική. Πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από πείνα. Το, ο αριθμός αυτός ανέβηκε σε 239 εκατομμύρια, δηλαδή 30% του πληθυσμού της Αφρικής. Από το 2002 μέχρι το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησε ε, κονδύλια ύψους ε, πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ για επιστημιστική βοήθεια στην υποσαχαρία Αφρική μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, το οποίο είναι το κύριο πλαίσιο για συνεργασία για την επιστημιστική ασφάλεια στην υποσαχαρία Αφρική. Επίση, υπάρχουν τρία ε, μέσα προέρχονται από τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο είναι ο προπολογισμό για την επιστημιστική ασφάλεια που διενεργεί παρεμβάσεις για βραχυπρόθεσμη βοήθεια, ε, μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση και τεχνική υποστήριξη για την επίτευξη επιστημιστική ασφάλεια ε, Με άλλα λόγια, παροχή σπόρων, εργαλείων και άλλων ε, αναγκαίων για την καλλιέργεια τροφίμων καθώς και μέσα αποθήκευσης. Έπειτα, το θεματικό πρόγραμμα για την επιστημιστική ασφάλεια που υποστηρίζει μεταξύ άλλων την έρευνα και την τεχνολογία για τη γεωργία και την βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και του οικοσυστήματος. Έπειτα, το 2008 δημιουργήθηκε το Food Facility για να, έχει, για να παρέχει μία άμεση βοήθεια σε επιστημιστικές κρίσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Πρωτού προχωρήσω στα κύρια βρήματα και τα συμπεράσματα, θα σας πω δύο λόγια για τον έλεγχο, το ελεκτικό συνέδριο ανέλησε το εάν η, η αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αφορά τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες και αν είναι αποδοτική. Εστιάσαμε <clears throat> στην άμεση υποστήριξη για την επισητιστική ασφάλεια, την πρόσβαση στα τρόφιμα και την ε, χρησιμοποίηση της βοήθειας αυτής. Έγιναν επιτόπιες επισκέψεις σε τρεις χώρες, την Αιθιοπία, το Μαλάουι και τη Ρουάντα. Έγινε επίσης μια έκθεση πιστοποίησης για άλλες χώρες. Θα ήθελα τώρα να αναφέρω τα κύρια ευρήματα και τα συμπεράσματα σματά του ελέγχου. Το συμπέρασμα είναι ότι η αναπτυξιακή βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την επισκεπτιστική ασφάλεια στην υποσαχάρη Αφρική είναι ιδιαίτερα αποδοτική και συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη τη επισητιστική ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα διεθνή παράγοντα στην διασφάλιση επισητιστικής ασφάλεια για πολλέ χώρε τη υποσαχάριας Αφρική και παρέχει υποστήριξη όσον αφορά την ε, πρόσβαση στα τρόφιμα και την διαθεσιμότητα. Έχει άμεση σχέση με τις προτεραιότητες των χωρών αυτών και λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα μέσα. Το, μέσο, το μέσο συστάθηκε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και αποτελεί μια πρόσθετη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διασφάλιση της επιστημικής ασφάλειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι παρεμβάσεις ε, στο μεγαλύτερο βαθμό τους ε, πέτυχαν το στόχο τους. Ωστόσο, υπάρχει περιθώριο για σημαντική βελτίωση σε πολλούς τομείς. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστίασε την αναπτυξιακή βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες με που έχουν επισητιστική που έχουν ανάγκη για επισητιστική βοήθεια, ωστόσο οι ανάγκες αυτές παραμένουν. Το, μέσο, το επισητιστικό μέσο συστάθηκε για να αντιμετωπίσει την επισητιστική κρίση του 2007, βραχυπρόθεσμα δηλαδή, και όχι τη μακροπρόθεσμη επισητιστική κρίση που παραμένει. Το μέσο αυτό αντιμετωπίζει προβλήματα όπως αναφέρθηκε η πρόσβαση στα τρόφιμα και η διαθεσιμότητα των τροφίνων. Δεν έχει δοθεί όμως αρκετή έμφαση στην σωστή διατροφή. Οι παρεμβάσεις πολλές φορές δεν θέτουν ξεκαθαρούς στόχους και ορισμένες φορές, για παράδειγμα στην ε, περίπτωση ΜΚΟ, δεν καταφέρνουν να επιτύχουν 100% τον στόχο τους. Μόνο οι μισές από τις ε, δράσεις στοχεύουν σε μακροπρόθεσμη αηφορία. Υπάρχουν επίσης μερικές ε, συστάσεις που το συνέδριο έχει κάνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Υπηρεσία ε, Εξωτερικής Δράσης. Για την προγραμματική περίοδο μετά το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να διεξάγουν μια αξιολόγηση της επιστημιστικής ε, κατάστασης στην υποσαχάρια Αφρική και να εξετάσουν τις ε, δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να εξετάσουν μαζί με άλλους εταίρους ενδεχομένω την βιωσιμότητα της χρηματοδότησης ε, επιγόντων και πρόσθετων μέτρων που ενδέχεται να χρειαστούν για να αντιμετωπίσουν πιθανές ε, μελλοντικές επισητιστικές κρίσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης της Ένωσης θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην επαρκή διατροφή, ενισχύοντας την συνεργασία, εντοπίζοντας και σχεδιάζοντας παρεμβάσεις και χρησιμοποιώντας τον ε, ε, διάλογο στα, ιδιαίτερα στο μέσο των ε, προγραμμάτων του προϋπολογισμού. Οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι στοχευμένες και μετρήσιμες με συγκεκριμένους δείκτες. Και τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι καλύτερα μετά και βασισμένα σε διεξοδικού ελέγχους και εκθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υποστηρίξει καλύτερα την βιωσιμότητα της καλλιέργεια και των κοινωνικών προγραμμάτων, διότι με τον τρόπο αυτό θα δοθεί περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη αποδοτικής γεωργίας και ανάλογων υπηρεσιών, υποδομών και θα διασφαλίσει ότι τα προγράμματα κοινωνικής μετάβασης θα παρέχουν επαρκή υποστήριξη στην ανάπτυξη των ε, δυνατοτήτων εισοδήματος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βέσπερ, για αυτήν την σύνοψη της ειδική έκθεσης. Τώρα ο εισηγητής Μπαρτστάς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πριν από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Βάισπερκ αλλά και όλη την ομάδα του. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη έκθεση, πολύ συγκεκριμένη, πολύ ακριβής και η οποία μας δείχνει ορισμένους δείκτες παρέμβασης, ε, ορισμένες ε, άγουσες που μπορούμε να ακολουθήσουμε δεν θα πρέπει να παραμείνει νεκρό γράμμα, θα πρέπει να εφαρμοστεί στην πράξη, εκεί που υπάρχουν κενά. Και χαίρομαι διότι στην Επιτροπή για τη Συνεργασία και την Ανάπτυξη ο κύριος Βάισμαν παρουσίασε την έκθεσή του χθες. Εγώ είμαι αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής για τη Συνεργασία για την Ανάπτυξη και νομίζω ότι είναι πολύ καλό το ότι παρουσιάζονται τέτοιες εκθέσεις ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Είναι καλό λοιπόν οι βουλευτές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα να είναι ενήμεροι και να μπορούν να αντλήσουν τα διδάγματα από όλες τις διαθέσιμες εκθέσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτό λοιπόν. Πιστεύω ότι βασικό συμπέρασμα της έκθεσής σας είναι ότι η αναπτυξιακή βοήθεια για την Αφρική και στην υποσαχάρη Αφρική είναι καλή, αλλά πάντοτε μπορούμε να κάνουμε και κάτι παραπάνω και πάντοτε μπορούμε να τελειοποιήσουμε ορισμένα σημεία. Χαίρομαι διότι η επισητιστική ασφάλεια αποτελεί μέρος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό το ταμείο είναι εξαιρετικά σημαντικό για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ανθρώπων που υποφέρουν. Και ακούσατε και ε, τα αριθμητικά στοιχεία που ανέφερε ο ομιλητής. Ένα λεπτό ζήτημα και θέτω το ερώτημα ε, και στα κράτη-μέλη, τα οποία βεβαίως δεν εκπροσωπούνται εδώ αλλά και στην Επιτροπή είναι το εξή. Στο 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη έχουμε την επιστημιστική ασφάλεια, η γεωργία, αναπτύξη της υπαίθρου κτλ. Σε όλα αυτά επικεντρωνόμαστε λιγότερο από ότι στο 9ο. Και φαίνεται αυτό αντιφατικό ως προς τους στόχους που έχουμε θέσει σε διεθνές επίπεδο. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα στην επιστημιστική ασφάλεια. Είναι πολύ συγκεκριμένο το ερώτημα που ε, απευθύνω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και νομίζω ότι έχουμε εκπρόσωπο εδώ της Κομισιόν. Η σύσταση στο πλαίσιο της κατάρτισης στρατηγικών εγγράφων αναχώρα θα μας επιτρέψουν να επικεντρωθούμε περισσότερο στην επισητιστική ασφάλεια, θα δώσουμε περισσότερη προτεραιότητα σε αυτό το θέμα, ναι ή όχι και ποια είναι τα συμπεράσματα που βγάζετε εσείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Κατά τα λοιπά, πιστεύω ότι η έκθεση αναφέρει ξεκάθαρα ότι δεν μπορούμε εμείς να είμαστε ο μοναχικός καβαλάρης. Πρέπει να ε, ε, συνδεθούμε, να συνδέσουμε όλα αυτά τα πράγματα με άλλους τομείς, με, άλλους, ε, με άλλα πεδία, με άλλες πολιτικές. Έχουμε τη μεταρρύθμιση της γεωργικής πολιτικής, έχουμε την πρωτοβουλία για το Διεθνές Εμπόριο της Εκτελεστικής Επιτροπής μαζί με τον Επίτροπο, έχουμε πολιτική αναπτυξιακή για την ανάπτυξη, Έχουμε διάφορα λοιπόν. Ε, υπάρχει συνοχή μεταξύ τους, αναρωτιέμαι. Μήπως ε, μπορούμε Μήπως εντοπίζουμε από εδώ και από εκεί στοιχεία αντιφατικά μεταξύ τους, από τη μία πολιτική στην άλλη. Και ό,τι γράφεται επί χάρτου δεν τηρείται πάντοτε, ξέρετε. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τους δωρητές, με τους χορηγούς, με όσους ε, δραστηριοποιούνται επιτόπου γιατί αυτοί πραγματικά γνωρίζουν ε, την Ήπειρο αυτό, αυτή. Η Αφρική είναι μια Ήπειρος που έχει δυνατότητες αυτοτροφοδοσίας. Μπορεί να θρέψει τον εαυτό της και όχι μόνο τον εαυτό της αλλά και άλλες περιοχές του κόσμου. Πολύ συχνά επιτόπου η κατάσταση είναι πολύ διαφορετική. Πολύ συχνά ε, διάφορες περιοχές της Αφρικής μαστίζονται από, πολέμους και συγκρούσεις. Επίσης διαπιστώνεται έλλειψη υποδομών και έλλειψη δυνατοτήτων αποθήκευσης. Μπορεί να γίνεται συγκομιδή, να μαζεύεται εισοδιά και τελικά να σαπίζει γιατί δεν μπορεί να βρει τα σωστά κανάλια για να διοχετευτεί στις αγορές και να μπορέσει και ο τοπικός πληθυσμός να τα αγοράσει και να τα καταναλώσει στη συνέχεια μια, ένα άλλο συμπέρασμα αυτής της ιδιαίτερης πραγματικά έκθεσης είναι κάτι το οποίο με ανησυχεί και έχει να κάνει με ε, το επισητιστικό μέσο 2008-2010. Μεταξύ αυτού και του νέου ταμείου που θα ξεκινήσει το 2014 υπάρχει ένα κενό. Και αυτό το κενό με ανησυχεί. Διότι διαπιστώνουμε ότι οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται όλο και περισσότερο, η προσφορά ποικίλει αναλόγως με την περίοδο, επομένως όλα αυτά έχουν άμεση συνέπεια στον, στην ανθρώπινη ζωή. Πώς θα ε, ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς, ε, πώς θα ε, ανταποκριθεί σε αυτό το ευμετάβολο, σε αυτή την τόσο διαφορετική και γρήγορη αλλαγή των τιμών και πώς θα την αντισταθμίσουμε αυτή την ε, μεταβλητότητα. Κάτι που μας ανησυχεί επίσης πάρα πολύ και ε, είναι μέρος των συμπερασμάτων των, της έκθεσης είναι το γεγονός ότι τα προγράμματα τελειώνουν και ποια συνέχεια θα δίδεται σε όλα αυτά. Μπορεί να επιτυχάνονται οι στόχοι, αλλά μετά να μην υπάρχει χρηματοδότηση και να μην συνεχίζεται το πρόγραμμα. Δηλαδή είναι σαν να σκοράρουμε ξαφνικά ε, και μετά να μένουμε άσφεροι. Νομίζω λοιπόν ότι η ποιότητα ε, μπορούμε να την εγγυηθούμε μόνο όταν εγγυόμαστε την συνέχεια σε όλα αυτά. Διαβάζω τα αποτελέσματα και βλέπω ότι οι στόχοι που έχουμε θέσει θα πρέπει να είναι πιο μετρήσιμοι και να έχουμε πιο συγκεκριμένα εργαλεία μέτρησης. Κατά τα λοιπά, συμφωνώ πολύ με τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, οι οποίες ε, περιγράφονται με πολύ αναλυτικό τρόπο και θα ζητούσα, θέλω να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να απαντήσει ε, στα διάφορα σχόλιά μου. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευχαριστούμε πολύ τον εισηγητή. Έχω λοιπόν δύο συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Καταρχήν η κυρία Ματιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή του ελεγκτικού συνεδρίου για την πολύ περιεκτική ανάλυση της κατάστασης και για τον πολύ θετικό απολογισμό που κάνει, παρόλο που επιδέχεται βελτιώσεων. Στην τρίτη παράγραφο του σχεδίου έκθεσης, στην πρώτη παρατήρηση του ελεγκτικού συνεδρίου, υπάρχει κάτι το ε, παράδοξο. Λέει ότι Κατά την κατάρτιση συνεργασιών, ε, στρατηγικών ε, συνεργασίας, η Επιτροπή δεν έλαβε πολύ υπόψη της κτλ. Και δεύτερον, έλλειψη προτεραιότητας στο πλαίσιο για, την, ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη. Η άποψη αυτή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επιτρέπει να αναλύσουμε τη λειτουργία του μέσου αυτού αλλά και τη διάρθρωση του μεταξύ των διαφόρων μέσων και εργαλείων για το ίδιο πεδίο δράσης ότι η παράγραφος 20 επισημαίνει ένα αδύναμο σημείο. Συμπληρωματικότητα των γραμμών του προπολογισμού, επιστημιστική ασφάλεια, ε, θέματα πόρων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Για την ίδια περίοδο διάφορα κράτη εποφελήθηκαν από δύο χρωματοδοτικά εργαλεία ε, και όχι από ένα. Μπορεί η Επιτροπή να μας εξηγήσει ε, ποια μεθοδολογία έχει ακολουθήσει. Ως προς το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ανάπτυξη, την ανάπτυξη η ανάπτυξη υπαίθρου και η επισητιστική ασφάλεια ήταν οι τομής προτεραιότητας για 17 χώρες για την περίοδο 96-2010 και για 12 χώρες για την περίοδο 2007-2013. Επομένως, η Επισητιστική ασφάλεια δεν ήταν τελικά η προτεραιότητα. Ενώ είναι στις πρώτες θέσεις του στόχους της χιλιετίας, αλλά είναι και στις πρώτες θέσεις στην ε, ε, ε, ε, της ανακοίνωσης της Επιτροπής του Μαρτίου του 2010. Έχουμε λοιπόν επικεντρωθεί και σε άλλους τομείς εκτός από την πείνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επισητιστική ασφάλεια που τελικά είναι ο φτωχός συγγενής της γενικότερη στρατηγικής για την ανάπτυξη. Μπορεί η Κομισιόν να μας εξηγήσει καλύτερα τι θα μπορούσε να έχει γίνει ώστε πιο συστηματικά να τοπίζουμε το θέμα της επιστημιστικής ασφάλειας. Πώς επιλέγονται οι τομείς προτεραιότητας. Πώς θα ληφθεί υπόψη η επιστημιστική ασφάλεια στην προγραμματική περίοδο μετά το 2013. Αυτό το καθήκον θα ανατεθεί σε άλλους δωρητές. Και για να ολοκληρώσω με κάτι το θετικό, Να σας πω ότι θέλει ένα πολύ καλό βαθμό ε, στην ε, έκθεση της, ε, του ελεκτικού συνεδρίου για τη Ρουάντα, την Αιθιοπία και το Μαλάου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τόιρ εξαφανίστηκε. Θα το διαπιστώσετε όλοι. Εγώ λοιπόν, είμαι Εγώ, λοιπόν τώρα θα είμαι πρόεδρος της συνεδρίασης και εισηγητής. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό. Ο κύριος Αντί. Ναι, Εν συντομία, λυπούμε, διότι δεν γίνεται αναφορά στο συντονισμό με τα κράτη-μέλη. Η ανάπτυξη είναι μέρος ε, των πολιτικών για να είναι κανείς χρήσιμος. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται αναφορά στο συντονισμό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμα και με τα Εθνικά Κοινοβούλιο. Το ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να εξετάσει συνολικά την παρέμβαση, την ευρωπαϊκή γίνεται λόγος μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην έκθεση αυτή. Λες και δεν υπήρχε τίποτα άλλο ή λες και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Εκφράζω ότι λύπη μου γι' αυτό. Θα πρέπει να συνηθίσουμε να μιλούμε πάντοτε ε, για τον συντονισμό με τα κρατημέλη, διότι τα κρατημέλη είναι αυτά που δαπανούν πάρα πολύ σημαντικά ποσά. Ευχαριστώ η κυρία Γκρέσλε. Εκτός και αν υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να παρέμβει, όχι. Η κυρία Κρεσλής και τελευταία. Ευχαριστώ πολύ, Μπάρτ. Κοίταξε, έχεις απόλυτα δίκιο. Πράγματι, είναι μια λεπτομερής έκθεση που μας προσφέρει πάρα πολλές πληροφορίες. Όμως η έκθεση δεν λέει βέβαια πώς ακριβώς θα ξεφύγουμε από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουμε εμπλακεί. Κάτι το οποίο έχουμε συνειδητοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ασκείται κριτική για το ότι δεν υπάρχουν οι σωστοί στόχοι, δεν ε, σημειώνεται επιτυχία. Τίθεται λοιπόν το εξή ερώτημα. Και τώρα τι θα κάνουμε. Ε, έχουμε διαθέσει τόσα πολλά κονδύλια και η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται. Εγώ λοιπόν δεν είμαι ευχαριστημένη και θα ήθελα να παρακαλέσω το ελεγκτικό συνέδριο να τοποθετηθεί, να μας πει ε, πώς θα αλλάξει την κατεύθυνση. Και έχεις δίκιο Μπάρτ, όσο δεν ανοίγουμε τις αγορές, απλά θα μπορούμε να μοιράζουμε ελεημοσύνη, αλλά δεν θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Για μένα είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Άρα δηλαδή με αυτά που έχουν κατατεθεί ως προτάσεις δεν είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη. Νομίζω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο και να βρούμε και άλλες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ασκήθηκε κριτική από αυτά που μας είπατε. Ήταν σαφές αυτό. Ο κ. Χάρκεν νομίζω είναι στην αίθουσα από πλευρά τη Επιτροπής για να υπερασπιστεί την άποψη της Επιτροπής και έχετε και το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω δύο λόγια για την κατάσταση της επισητιστικής ασφάλειας και για τις εξελίξεις από τότε που ε, δημοσίευσε την έκθεσή του το ελεγκτικό συνέδριο. Από τη δημοσίευση λοιπόν της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέχισε να υποστηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες επισητιστικής ασφάλειας για να αντιμετωπίσει τις επισητιστικές κρίσεις στην Αφρική και μάλιστα στην υποσαχάρια Αφρική. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, οι τιμές πράγματι συνεχίζουν να διαταράσσουν την επισητιστική ασφάλεια. Υπογραμμίζουμε ότι το ελεκτικό συνέδριο έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά. Η Επιτροπή πράγματι ε, συμφωνεί με την πλειονότητα των διαπιστώσεων της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου και βασιζόμαστε στην έκθεση αυτή για να επιταχύνουμε την ε, εφαρμογή διαφόρων μέτρων. Και αυτή τη στιγμή ε, βρισκόμαστε σε φάση η εφαρμογής και υλοποίησης των συστάσεών μας. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια σημεία που αναφέρατε. Πρώτον, η σημασία της επισητιστικής ασφάλειας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας και στο πλαίσιο της βοήθειας της Ευρώπης για την ανάπτυξη. Πράγματι, μπορεί κανείς να εκφράσει τη λύπη του, διότι ε, διαπιστώσαμε μία υπαναχώρηση στον αριθμό των χωρών που επέλεξαν την επισητιστική ασφάλεια ως βασικό πυρήνα για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές τους πριν και μετά το 2010. Ως, σε ορισμένα γεωγραφικά μέσα το είδαμε αυτό. Και θα δούμε το περιθώριο που έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τούτων λεχθέντων, παρά την κατάσταση αυτή, διαπιστώνουμε με τις εκθέσεις που συντάσσουμε το πλαίσιο της ε, ε, πρωτοβουλία για την επιστημιστική ασφάλεια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο πρώτος δότης, ο πρώτος εγγυητής αν θέλετε ε, για την επιστημιστική ασφάλεια περισσότερο και από τις Ηνωμένε Πολιτείε και αυτό δεν είναι διόλου αμεληταίο. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σχολιάσω ορισμένα ζητήματα. Τον τρόπο με τον οποίο προτιθέμεθα να υλοποιήσουμε αυτές τις συστάσεις. Πρώτον, πώς θα λάβουμε υπόψη μας την επισητιστική ασφάλεια στις δημοσιονομικές προοπτικές για το 2014 μέχρι και το 2020. Το ελεκτικό συνέδριο προτείνει να έχουμε μια πιο καλά δομημένη ανάλυση είναι κάτι το οποίο συμμεριζόμαστε εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πράγματι θα αναλύσουμε την κατάσταση όλων των χωρών σε φάση ανάπτυξης, των αναπτυσσόμενων χωρών, για να δούμε ε, ποιες πάσχουν από χρόνια επισητιστική ασφάλεια. Επί τη βάση λοιπόν 50 δικτών περίπου, περίπου ε, έχουμε εντοπίσει αυτές τις χώρες 52 χώρες, δεν ξέρω αν τις βλέπετε με κόκκινο χρώμα στο χαρτί που σας δείχνω, δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα και μπορείτε να το δείτε στις οθόνες σας. Ο Γενικός Διευθυντής της Europe Ed και ο κύριος Σίτιφαν που είναι CEO του ΟΕΣ κάλεσαν τους επικεφαλείς αντιπροσωπιών να ξεκινήσουν ένα πολιτικό διάλογο με τις χώρες αυτές, ώστε και οι χώρες αλλά και οι δωρητές να λάβουν υπόψη τους αυτή την κατάσταση της χρόνιας έλλειψης επισητιστικής ασφάλειας. Δηλαδή της χρόνιας ανεπάρκειας τροφίμων. Μπορούμε λοιπόν να διαπιστώσουμε ότι πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδειξε ότι είναι ικανή να αντιμετωπίσει τις επισητιστικές κρίσεις, κινητοποιώντας με την υποστήριξη των δημοσιονομικών αρχών πολύ σημαντικά ποσά. Εάν δούμε το food facility, το μέσο αυτό για τα τρόφιμα, το επισητιστικό, μπορούμε πράγματι να εκφράσουμε την ικανοποίησή μας για την ταχύτητα της αντίδρασής μας, για την ταχύτητα της ανταπόκρισής μας και της εφαρμογής όλων αυτών των μέτρων. Και βέβαια όλα αυτά τα κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες της επισητιστικής κρίσης. Βοηθούμε τις πιο ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες να ε, ξεπεράσουν αυτή την κρίση και να μπορέσουν να συνεχίσουν στη συνέχεια. Εξού και πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να δώσει περισσότερη έμφαση στις αιτίες που προκαλούν επισητιστική κρίση. Ε, και αυτό ήταν και η βάση της κατάρτισης της νέας πολιτικής που επικύρωσε το Σώμα των Επιτρόπων στις 3 Οκτωβρίου, που είναι η πολιτική της επιμονής. Αντίσταση. Σκοπός είναι σε κάθε κλίμακα σε κάθε επίπεδο να μπορεί ο κάθε ένας να αντέξει, ο κάθε, το κάθε ε, φορέας ε, να μπορέσει να αντέξει και να ξεπεράσει την κρίση σε επίπεδο νοικοκυριού, τοπικής κοινότητας, παραπάνω παραπάνω. Ε, και μπορούμε να έχουμε παραδείγματα που μας ενθαρρύνουν. Ο Νίγηρας, η χώρα που επλήγει περισσότερο από την κρίση του Σαχέμ. Και χάρη σε μια εξαιρετικά βολονταριστική πολιτική είναι η χώρα που αντιμετωπίσε ε, καλύτερα από όλες τις άλλες την κρίση. Ε, υιοθέτησε μέτρα παρέμβασης και έτσι με τους δικούς, του, δικούς της πόρους η χώρα αυτή μπόρεσε να αντιμετωπίσει την κρίση. Κάτι που αναφέρθηκε επίσης είναι η αναγκαία ε, συνεργασία, ο αναγκαίος συντονισμός με τους δωρητές. Πράγματι είναι αυτό πολύ σημαντικό. Ε, συμφωνούν επ' αυτού και οι υπηρεσίε για την αναπτυξιακή βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, συμφωνούν και οι χώρες του Συμβουλίου που ε, έχουν έδρα στο ΚΟΝΤΕΒ. Και πράγματι υπάρχουν δωρητές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, όχι απαραίτητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά άλλοι. Θέλω τώρα να επανέλθω στο θέμα του ιδιωτικού τομέα της αγοράς, των αγορών και της διατροφής και του υποσυτισμού. Ο παιδικός υποσυτισμός είναι πράγματι ένα πρόβλημα το οποίο γνωρίζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά τελικά δεν το γνωρίζουμε πολύ καλά. Η έκθεση του 2008 που είναι η πιο ενδελεχής επιστημονική έκθεση ε, ιατρικής έρευνας κατέδειξε πόσο καταστροφικός είναι ο χρόνιος υποσυτισμός. Αυτό το οποίο υποφέρει και παθαίνει δηλαδή ένα παιδί που πάσχει από υποσυτισμό είναι ε, κάτι το φοβερό και ε, φαίνεται ακόμα και όταν σταματήσει. Δηλαδή ένα παιδί που ε, είχε χρόνιο υποσυτισμό έχει μετά προβλήματα υγείας παρόλο που μπορεί να έχει σταματήσει ο υποσυτισμός του και δεν έχει εξόψεως την εικόνα που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην τηλεόραση. Σε κάθε περίπτωση 3,5 εκατομμύρια παιδιά που υποσυντητίζονται πεθαίνουν κάθε χρόνο. Αυτό είναι ένα νούμερο ανατρεχιαστικό. Και το επίσης εξαιρετικά αρνητικό είναι ότι αυτά που τελικά επιζούν τα παιδιά ε, δεν πρόκειται να αναπτυχθούν ε, βάσει των δυνατοτήτων τους. Δηλαδή ο χρόνιος υποσυντισμός ο χρόνιος υποσυτισμός αφήνει, ε, καταφέρνει ανεπανόρθωτο πλήγμα στην ψυχική, νοητική, πνευματική, σωματική ανάπτυξη του παιδιού. Έχουμε προβληματιστεί πολύ για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το αυτό το θέμα παγκοσμίω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. να Έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία πολύ συγκεκριμένη και ο Επίτροπος Πίμπαλς είναι εξαιρετικά δραστήριος. Είναι μέλος της ομάδας των 25 ατόμων που ηγούνται αυτής της πρωτοβουλίας, παρέστη στη Σύνοδο του Λονδίνου για την πείνα, την καταπολέμηση ε, της πείνας, φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να σώσουμε 7 εκατομμύρια παιδιά που πάσχουν από χρόνιο υποσυτισμό από σήμερα μέχρι το 2022. Ο Επίτροπος Πίμπαλς ήταν εξαιρετικά σαφής, δεν θέλει να αφήσει στο διάδοχό του το θέμα αυτό και μας ζήτησε να επανέλθουμε με πολύ συγκεκριμένο και λεπτομερές σχέδιο. Δεύτερον, πρέπει να συνεργαστούμε στενά με τον ιδιωτικό τομέα, στην άτυπη ή στην επίσημη μορφή του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη γεωργική για την αγροτική παραγωγή σε αυτές τις χώρες. Στην Αφρική, το μέρος τον, το ποσοστό των τροφίμων που καταναλώνουν οι Αφρικανοί ε, πέφτει ραγδαία. Εισάγουν πλέον το 30% των αναγκών τους. Ό,τι παράγουν ε, το καταναλώνουν όλο και λιγότερο. Περίπου 28 δις δολάρια σε εισαγωγές λοιπόν ετησίως. Είναι απαραίτητο να αυξηθεί η αγροτική δραστηριότητα στην Αφρική, να ενισχυθεί, να δώσουμε ε, στήριξη στις χώρες για γεωργική πολιτική πολύ καλύτερα προκαθορισμένη. Όλα αυτά αφορούν και τους μικρούς αγρότες, τους μικρούς καλλιεργητές για να ενταχθούν καλύτερα στην αλυσίδα αξιών της ιδιωτικής αγοράς. Πρόσβαση στην αγορά, σωτιά, απώλειες, αντισταθμίσεις, διάδραση και συνεργασία με τα κανάλια της αγοράς. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Τέλος, κάτι που ε, ανέφερε η κυρία Ματιού. Διάρθρωση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Ανάπτυξη και του ε, Ταμείου ε, FSTP. Σήμερα, ε, οι θεματικοί άξονες στρέφονται γύρω από συγκεκριμένα σημεία, δηλαδή ενίσχυση του δημόσιο αγαθού παγκοσμίω. Π.χ. η έρευνα για θέματα αγροτικά, γεωργικά. Αυτό δεν θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από συγκεκριμένου μόνο εις βάρος άλλων από τη στιγμή που τα ωφέλη θα είναι για όλον τον κόσμο. Για να αντιμετωπίσουμε τις επισητιστικές κρίσεις ε, ε, τις οποίες δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τα κλασικά γεωγραφικά μέσα, γι' αυτό έχουμε ε, δημιουργήσει αυτό το ταμείο, το FSTP και έχουμε το νέο πρόγραμμα το παγκόσμιο κοινό αγαθό, δημόσιο αγαθό και προκλήσεις. Και εκεί έχουμε το θεματικό πρόγραμμα επισητιστική ασφάλεια, ενδεχομένως στη θέση των γεωγραφικών μέσων. Θα έπρεπε να είχαμε τα γεωγραφικό αμέσα, θα διορθώσουμε ε, αυτή την αδυναμία. Ελπίζω και πιστεύω ότι απάντησα στις ερωτήσεις που μου έχετε θέσει. Ευχαρίστω ε, να ξαναπάρω το λόγο. Είμαι στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ωραία λοιπόν. Ε, ακούσαμε πάρα πολλές ε, πληροφορίες, επίσης μπορούμε και να χρησιμοποιήσουμε. Η έκθεση μπορεί και να τροποποιηθεί. Έχουμε χρόνο μέχρι τις 14 ε, Οκτωβρίου. Οι πληροφορίες που μας ε, καταθέσατε είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που θέλει να προσθέσει κάτι. Μήπως το λεκτικό συνέδριο, ο κύριος Βέσμπερκ, μήπως ε, επιθυμείτε εσείς να τοποθετηθείτε. Ο κύριος Βέσμπερκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λίγα λόγια θα πω. Έγινε ένα σχόλιο για το κατά πόσο πρέπει να δούμε λιγάκι ή αν είδαμε ε, το θέμα του συντονισμού των δωρητών. Αναφέρεται ε, αυτό το θέμα σελίδα υπαριθμών 24. Δεν το είπα εγώ προφορικά, αλλά πρέπει να πω ότι δεν είναι αρκετός, δεν είναι ικανοποιητικός ο συντονισμός για να επιτευχθούν οι στόχοι. Επίση, σε τέτοιο ερώτημα κατά πόσο έχουμε να υποβάλουμε περαιτέρω συστάσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά μας. Κοιτάξτε, δεν έχουμε περαιτέρω συστάσεις πέρα από τις πέντε οι οποίες αναφέρονται στην έκθεση. Και θέλω να πω, όπως όλοι σας πολύ καλά γνωρίζετε, αυτήν την ειδική έκθεση ε, προσπαθούμε να την κρατήσουμε ε, όσο περισσότερο, όσο πιο στοχευμένοι μπορούμε. Στοχευμένοι σε συγκεκριμένα θέματα. Ε, δεν μπορούμε να τα θίξουμε όλα. Έχουμε πέντε συγκεκριμένες συστάσεις στις οποίες έχουμε καταλήξει και νομίζω ότι η δική μας στάση θα συμβάλλει στο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα. Πρόεδρος, ε, πολύ ωραία. Ας το κλείσουμε λοιπόν ε, το θέμα εδώ. Ε, το θέμα σίγουρα χρήζει ακόμα της προσοχής μας. Αλλά κοιτάξτε, επειδή τώρα έχω και την ιδιότητα του Προέδρου, ε, πρέπει να μην ξεχνάμε και το χρόνο που τρέχει. Ήδη είμαστε ε, καθυστερημένοι κατά ένα τέταρτο. Ευχαριστώ λοιπόν όλους τους συναδέλφους ε, που έλαβαν το λόγο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ελληνικό Συνέδριο. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου για να καταθέσουμε τις τροπολογίες, δηλαδή μέχρι την επόμενη Δευτέρα 12 η ώρα. Έτσι λοιπόν ε, κλείνει το σημείο υπαριθμών 9 της ημερήσιας διάταξης και πάμε στο 10 που είναι μια μελέτη με θέμα ο ρόλος της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Έχουμε εδώ τους καλεσμένους ε, που συνέταξαν την έκθεση Μάρκους Σμιτ και Ιρένε Στεμπράιν. Ε, οι δύο μπορούν να έρθουν αν θέλουν εδώ. Όχι, ε, θα κάτσουν στη θέση τους. Ωραία, μείνετε εκεί. Ε, εγώ σας ε, γνωρίζω βέβαια γιατί εγώ ήμουν ο εισηγητής που παρακολούθησε και αυτός τη μελέτη. Έχουμε δύο συνεργάτες του Ταμείου Πασκάλ Ντεγκρούς Εσείς, σε εσά κατακυρώθηκε η μελέτη και αυτό λόγω της ποιότητας που σας ε, χαρακτηρίζει. Και θα ήθελα να ευχαριστώ και τον κύριο Χέλμουτ Βέρνα, ο οποίος ε, παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς αυτή τη μελέτη. Αυτή λοιπόν η μελέτη εξετάστηκε εξονυχιστικά. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Βέρνα, κάλεσε μένα και άλλους επανειλημμένα να συμπεριλάβουμε κάποια στοιχεία στην έκθεση αυτή. Στην έκθεση λοιπόν, στη μελέτη, επανέρχομαι σε μία παράκληση, παλαιότερη δική μου. Τότε λοιπόν είχα διαβάσει σε, μία, σε ένα άρθρο της Μαρτίνα Κοβακιόβα από την Σλοβακία, είχε γράψει ένα άρθρο η δημοσιογράφος αυτή σχετικά με την απάτη με κονδύλια του κοινωνικού, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και μετά αυτή απολύθηκε. Σκέφτηκα λοιπόν ότι η ερευνητική ε, δημοσιογραφία είναι πολύ σημαντική κυρίως σε περίοδους κρίσης. Εδώ τίθεται θέμα εμπιστοσύνη. Οι άνθρωποι έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους ε, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε λοιπόν θεματοφύλακες. Ποιοι μπορούν να επαγρυπνούν, καταρχήν οι πολιτικοί. Εμείς ε, θα πρέπει να είμαστε οι ε, άγρυπνοι φύλακες οι whistleblowers, οι πληροφοριοδότες, οι δικαστές ε, αλλά και οι δημοσιογράφοι έχουν ακριβώς αυτή την ε, αποστολή του άγρυπνου φύλακα οι οποίοι οι ε, δημοσιογράφοι έχουν την ε, ευθύνη ή την αρμοδιότητα ε, να ερευνήσουν θέματα. Αντιμετωπίζουν όμως πολλές φορές εμπόδια. Εμπόδια από τους ε, αρχισυντάκτες τους. Πολλές φορές λένε «Μα δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχουν χρήματα». Τίθεται λοιπόν πολύ συχνά το ερώτημα και εγώ που θα τις βρω τις απαραίτητες πληροφορίες. Κατόπιν πολλές φορές υπάρχει το εμπόδιο εξακρίβωσης της πληροφορίας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ε, ως Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμών αποφασίσαμε να χρηματοδοτήσουμε αυτή τη μελέτη, να δώσουμε τη δυνατότητα ε, να παρακολουθηθεί η εργασία αυτών των δημοσιογράφων για έξι ε, ολόκληρους μήνες. Ο Μάρκο, όχι, η κυρία Σμιτ παίρνει το λόγο και λέει θα κάνω την παρουσίασή μου στα αγγλικά γιατί η μελέτη είναι στα αγγλικά. Εδώ αντιπροσωπεύω περίπου 100 δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη, οι οποίοι με βοήθησαν σε αυτή τη μελέτη. Και οι τελευταίοι έξι μήνες ήταν για μένα μία επιβεβαίωση του ότι το δημοσιογραφικό δίκτυο, έτσι όπως ε, αναδύεται το δημοσιογραφικό δίκτυο ε, των ερευνητικών δημοσιογράφων, έχει αποτελέσματα. Αυτή η μελέτη δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη βοήθεια πάνω από 100 δημοσιογράφων σε όλη την Ευρώπη. Και θα σας κάνω μια σύντομη παρουσίαση, θα σας δείξω μερικές διαφάνειες και θα απαντήσω σε ενδεχομένες ερωτήσεις και ελπίζω πληροφορίες αυτές να χρησιμοποιηθούν με καλό τρόπο, διότι οι δημοσιογράφοι έχουν την ανάγκη της βοήθειάς μας. Επί έξι μήνες εργαστήκαμε σε αυτή τη μελέτη, στόχος της οποίας όταν κερδίσαμε τον ε, διαγωνισμό ήταν να ανακαλύψουμε το εάν η ερευνητική δημοσιογραφία μπορεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση της απάτης με τα ευρωπαϊκά κονδύλια και μπορούμε να πούμε ότι βοήθησε κάπως μέχρι τώρα. Μένουν πολλά όμως ακόμα που μπορούν να γίνουν. Εμείς εστιάσαμε σε αυτά που, μπορεί, που μπορούν να γίνουν. Προσπαθήσαμε να εστιάσουμε στις βελτίστες πρακτικές που ισχύουν μέχρι τώρα και όχι σε αυτά που δεν λειτουργούν. Γιατί πολλές φορές δεν λειτουργούν πολλά πράγματα. Δημιουργήσαμε μερικέ συστάσεις τις οποίες δεν απευθύνουμε άμεσα προς τα ευρωπαϊκά όργανα ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι πιστεύουμε ότι ο ίδιος ο δημοσιογραφικός κλάδος χρήζει αναδιάρθρωσης. Εμείς ως δημοσιογράφοι γνωρίζουμε ότι δεν λαμβάνουμε κριτική από εξωτερικούς φορείς με καλό τρόπο. Προτιμούμε ίδιοι να ασκούμε κριτική στον εαυτό μας. Εν συντομία θα σας πω τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Αποφασίσαμε να απεικονίσουμε το ερευνητικό τοπίο στο 2007 έτσι ώστε να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε το πώς γίνεται η ερευνητική δημοσιογραφία. Αναλύσαμε και αξιολογήσαμε το ποσοστό της ερευνητικής δημοσιογραφίας όσον αφορά τις δαπάνες και τα εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να αναλύσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε και να κάνουμε συστάσεις και στα ευρωπαϊκά όργανα και στους ίδιους τους δημοσιογράφους για το πώς να αυξήσουν την επιρροή τους στην ερευνητική δημοσιογραφία. Εγώ ίδια είμαι ερευνητική δημοσιογράφος από τις κάτω χώρες, είμαι επικεφαλής της έρευνας και είμαι επικεφαλής της ε, φλαμανδόφωνης ε, κοινότητας ερευνητικών δημοσιογράφων. Εργάζομαι στο Ίδρυμα Pascal de στο Βέλγιο, το οποίο προωθεί την ερευνητική δημοσιογραφία στην φλαμανδόφωνη κοινότητα του Βελγίου Δίπλα μου είναι ο κύριος Δεμπράουν, είναι ο διευθυντής του ιδρύματό Πασκάλ Ντεγκρό. Αυτή η μελέτη δεν θα μπορούσε να γίνει χωρί την ερευνητική ομάδα μου. Η αποτελείται από έξι δημοσιογράφους. Θα βρείτε το όνομά τους στην έκθεση. Και η ομάδα αυτή ήταν, ε, είχε αποφασιστική σημασία στην έρευνα αυτή. Είχαμε συμβολές από 23 δημοσιογραφικές ε, ενώσεις στην Ευρώπη και είχαμε τη συνεισφορά 40 ανώνυμων και 37 επώνυμων δημοσιογράφων. Ορισμένοι δημοσιογράφοι δέχτηκαν να μας μιλήσουν μόνο ανώνυμα, διότι αυτά που μας είπαν ήταν πάρα πολύ σημαντικά και άσκησαν κριτική και για το ίδιο το επάγγελμά τους και για τα μέσα για τα οποία εργάζονται, αλλά και για τα ίδια τα ευρωπαϊκά όργανα και ορισμένοι από αυτούς τους δημοσιογράφους αισθάνθηκαν πιο ελεύθεροι μιλώντας ανώνυμα. Και αυτό συνδέεται και με αυτό που είπε ο κύριος στην ε, εισαγωγή του, ότι είναι πολύ δύσκολο να ασκήσουν δημοσιογράφοι κριτική για τα εκτενόμενα στην ίδια του τη χώρα. Προσπαθήσαμε λοιπόν να απεικονίσουμε την κατάσταση όσο το δυνατόν πληρέστερα και δώσαμε στους ε, δημοσιογράφους τη δυνατότητα να μιλήσουν ανώνυμα. Αρκετοί όμως από αυτούς δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να παραμείνουν στην ανωνυμία. Είχαμε λοιπόν εισφορά περίπου, στην εισφορά περίπου 50 οργανισμών, ε, ανάμεσα τους και το ελεκτικό συνέδριο και ε, διαφορετικές γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνομιλήσαμε με ανθρώπους από εκεί. Χρησιμοποίησαμε πάνω από 50 συνόψεις της, ε, σχετικές με το τοπίο, το δημοσιογραφικό τοπίο στην Ευρώπη. Δεν υπήρχε όμως κάποια συνολική θεώρηση του τοπίου της ερευνητικής δημοσιογραφίας και εμείς προσπαθήσαμε στο παράδειγμα 1 της ε, μελέτης να δώσουμε μια εικόνα της κατάστασης της ερευνητικής δημοσιογραφίας στην Ευρώπη. Επίσης, ε, μιλήσαμε σε πάνω από 40 δημοσιογράφους και υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να μελετήσουμε την κατάσταση εις βάθος. Χρειαστήκαμε καταρχάς έναν ορισμό της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Ακούγεται πιο εύκολο από ότι είναι στην πραγματικότητα. Τι είναι λοιπόν η ερευνητική δημοσιογραφία. Η προκήρυξη ήδη μας έδωσε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές. Δημοσιογραφία που ασκεί κριτική σε βάθος και δημιουργεί ειδήσει που δεν θα μπορούσαν να είχαν βγει προς το έξω χωρίς την δουλειά αυτή των ερευνητικών δημοσιογράφων. Δεν οφείλεται μόνο στην ε, πληροφόρηση για καινούργιε ειδήσει, αλλά και στην ε, διαφορετική με νέο τρόπο μετάδοση των πληροφοριών. Είτε με ποσοτικό ποιοτική έννοια, είτε με ποιοτική έννοια, είτε με ένα συνδυασμό και των δύο. Αυτό ο ορισμό χρησιμοποιείται από τον Σύνδεσμο Ερευνητικών Δημοσιογράφων για τον οποίο εργάζομαι τα τελευταία δέκα χρόνια και τίνει να γίνεται περισσότερο αποδεκτός ως ένας επίσημος ορισμός της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Και κύριο σημείο των προσπαθειών μας ήταν η κριτική και εις βάθος δημοσιογραφία, η οποία φέρνει στο φως νέα τα οποία δεν θα μπορούσε να φέρει στο φως χωρίς την ύπαρξή της. Και οι ειδήσει που ήρθαν στο φως σχετικά με την απάτη για τα ευρωπαϊκά κονδύλια δεν θα μπορούσαν να βρεθούν χωρίς την δουλειά αυτή των ερευνητικών δημοσιογράφων. Θα επανέλθω σε αυτά τα ρεπορτάζ. Ασχοληθήκαμε λοιπόν με τις περιπτώσεις απάτης ευρωπαϊκών κονδυλίων τα τελευταία πέντε χρόνια. Και δώσαμε προσοχή σε ειδήσει τις οποίες ανακάλυψαν οι δημοσιογράφοι. Θέλουμε, να σας δείξουμε αυτό που κατάφεραν και πώς οι δημοσιογράφοι μπορούν να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της απάτης παρά να δώσουμε βάρος σε ειδήσει που ήρθαν στο φως από άλλα όργανα. Για παράδειγμα από το ελεκτικό συνέδριο. Εμείς θέλουμε να δώσουμε προσοχή στο ρόλο των ερευνητικών δημοσιογράφων. Τι έχουμε λοιπόν. ερευνητικό ρεπορτάζ όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κονδύλια, δαπάνες και έσοδα. Ως δημοσιογράφοι δώσαμε βάρος στις δαπάνες. Ψάξαμε για αναφορέ ιδία πρωτοβουλία, όπω το λέμε. Μπορείτε να το δείτε στο παράρτημα 2 τη έκθεση. Αναλύσαμε ένα χρονικό περιθώριο 5 ετών. Πολλέ όμω από αυτέ τι ε, περιπτώσει ανάγονται πολύ ε, παλαιότερα. Κοιτάξαμε όλα τα μέσα ενημέρωσης, κοιτάξαμε βάσεις δεδομένων, ειδήσεων, είχαμε το συνεργασία με δίκτυο πάνω από 100 δημοσιογράφων σε όλη την Ευρώπη, σε πολλές γλώσσες και όχι μόνο σε ειδήσει ε, και πληροφορίες στα αγγλικά. Εξετάσαμε αναφορές από όλα τα 27 κράτη-μέλη έτσι ώστε να δούμε ποιες ειδήσει ήταν σημαντικές σε κάθε χώρα, στη δική σας χώρα, στη δική σας γλώσσα. Σε όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Και ως τη λύση, κάναμε έκκληση στη μνήμη των ανθρώπων, διότι πολλές φορές οι βάσει δεδομένων είναι προστατευμένε, είναι απόρριτε. Έχουμε παράδειγμα μιας χώρας όπου ένας ε, εκφωνητής ειδήσεων δεν επιτρέπεται να δημοσιεύει ειδήσει στην προσωπική του ιστοσελίδα, διότι θεωρείται ανταγωνισμός από, τις, ε, από τα έντυπα μέσα, από τις εφημερίδες. Πολλέ φορέ λοιπόν αντλήσαμε πληροφορίε από Μνήμα των δημοσιογράφων. Η έρευνα είναι αντιπροσωπευτική, ποιοτικά και όχι τόσο ποσοτικά. Και εάν μας διέφυγε κάποιο θέμα, ελπίζουμε να μας επιστήσουν την προσοχή σε αυτό οι συνάδελφοι. Και δημιουργήσαμε μία βάση δεδομένων με τις ειδήσει αυτές, έτσι ώστε οι δημοσιογράφοι στο μέλλον να μπορέσουν να ανατρέξουν σε αυτές και να τις ε, διερευνήσουν περαιτέρω. Διότι όπως προανέφερα η συνεργασία είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κάτι στο οποίο πρέπει να εργαστούμε όχι μόνο οι δημοσιογράφοι σε σχέση με τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και οι δημοσιογράφοι μεταξύ τους. Πρέπει να συνεχίσει ο ένας το έργο του άλλου έτσι ώστε να δώσουμε την καλύτερη και πληρέστερη δυνατή είδηση. Τι βρήκαμε λοιπόν από την βάση αυτή δεδομένων. Είχαμε πάνω από 230 πάνω από 233 θέματα σε 27 κρατη σε περίοδο 5 ετών. Τα, οι περισσότερες αυτές ε, ειδήσει προήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο. και μετά από ορισμένε χώρε οι οποίε μπορεί να μην είναι οι συνήθει ύποπτοι, για παράδειγμα η Γερμανία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία. Επίσης αρκετέ ε, ιστορίες προήλθαν από την Ισπανία. Όπως βλέπετε και στο διάγραμμα στην οθόνη σας. Πολλές από τις ε, χώρες αυτές, όπως για παράδειγμα οι σκανδιναβικές χώρες, Σουηδία και η Δανία, έχουν μακρά παράδοση στην ερευνητική δημοσιογραφία. Δεν θα τις δείτε όμως στο διάγραμμα. Όταν ψάξαμε για μια εξήγηση του φαινομένου, είδαμε ότι 233, ε, τα 233 θέματα μπορεί να ήταν λίγα, αλλά εάν κοιτάξουμε την ε, κατανομή αναχώρα θα δείτε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πάρα πολλέ. Σλοβακία, Βουλγαρία, Γερμανία αρκετέ, αλλά σε άλλες χώρες όπως για παράδειγμα στην Ιταλία δεν είχαμε σχεδόν καθόλου θέματα. Το θέμα ήταν, τα θέματα ήταν ενιαία. Ασχολούνταν κατά κύριο λόγο με την ε, κατάχρηση εξουσίας, από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως εσάς για παράδειγμα, αλλά και από μεμονωμένες εταιρείες ή από γενικούς διευθυντές εταιριών, από κατάχρηση εξουσίας από τα ευρωπαϊκά όργανα και από μεμονωμένα άτομα που εργάζονταν στα ευρωπαϊκά όργανα. Αυτά όλα μπορείτε να τα βρείτε στην έκθεση. Δεν είναι κάτι σπάνιο, συμβαίνει συχνά. Επίσης, ως δημοσιογράφοι μας αρέσει να διηγούμαστε ιστορίες. Χρειαζόμαστε έναν πρωταγωνιστή. Ένα όνομα. Γνωστό όνομα. Πολλές φορές αυτό που βρήκαμε, για παράδειγμα ένας δημοσιογράφος από το Ηνωμένο Βασίλειο μας είπε ότι αν ψάχνετε για κατάχρηση χρήματος, τότε χρειάζεστε ένα όνομα. Εάν βρείτε όνομα, τότε θα έχετε και την είδηση. Είχαμε λοιπόν πολλές περιπτώσεις τέτοιες. Είχαμε πάρα πολλές ε, περιπτώσεις για δαπάνες, πολύ λίγες για έσοδα και φαίνεται πως η απάτη σχετική, σχετική με τα έσοδα δεν είχε πολλές ειδήσει να δώσεις. Δεν θέλουμε όμως να εξάγουμε εκ των προτέρων συμπεράσματα. Όμως αυτό που βρήκαμε είναι πολλές περιπτώσεις απάτης σε δαπάνες, κυρίως με τις επιχορηγήσεις στη Γεωργία, στην Αλία και στα διαρθρωτικά ταμεία. Και αυτά υπήρχαν εκεί, διότι υπήρχαν ορισμένοι αποφασισμένοι δημοσιογράφοι, οι οποίοι ήταν αποφασισμένοι να διερευνήσουν, για παράδειγμα, τις ε, απάτες με τις γεωργικές επιχορηγήσεις. Η γεωργία είναι ένα τομέα ο οποίο απορροφά πάρα πολλά κονδύλια και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις κατάχρησης κονδυλίων. Και υπάρχει πολύ λίγος ε, έλεγχος στις ε, δαπάνες αυτών των κονδυλίων. Επίσης, κοιτάξαμε το μέγεθος των δημοσιεύσεων. Αλλά στη Γαλλία η ερευνητική δημοσιογραφία είναι πολύ μικρή κλίμακα. Επίσης, πολλές ειδήσει υπήρχαν στο διαδίκτυο, στην Ουγγαρία. Για παράδειγμα, η οποία είναι πρωτοπόρο στην ε, διαδικτυακή ερευνητική δημοσιογραφία. Και πολλές φορές οι δημοσιογράφοι εργάζονται αμυστή, εθελοντικά, δεν θα επανέλθω σε αυτό. Επίσης, προσπαθήσαμε προσπαθώντας να βρούμε τις ε, αιτίες που κρύβονται πίσω από αυτά τα φαινόμενα, κοιτάξαμε τις διάφορες τάσεις που επικρατούν και απευθυνθήκαμε στα μέσα, στα μέσα ενημέρωσης. Τους ρωτήσαμε γιατί δεν ασχολείστε ή κυρίως, δεν ασχολείστε με αυτά τα θέματα. Μας ανέφεραν ε, την οικονομική κρίση ως ε, δικαιολογία. Ωστόσο, εμείς ανακαλύψαμε ότι η απόφαση για ερευνητική δημοσιογραφία δεν βασίζεται μόνο σε οικονομικούς λόγους. Εξαρτάται από την θέληση ή όχι. Και αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με κάποιο θέμα το κάνουν ανεξάρτητα με το αν υπάρχουν οικονομικοί πόροι ή όχι. Μετά ρωτήσαμε εάν υπάρχει χώρος για ερευνητική δημοσιογραφία σε ένα δελτίο ειδήσεων. Έπειτα, οι δεξιότητες. Μπορούν οι δημοσιογράφοι να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Όχι, δεν μπορούν. Αυτό βρήκαμε, διότι δεν είναι πολλές φορές κατάλληλα καταρτισμένοι για ερευνητικό ρεπορτάζ. Επίσης, η πίεση παίζει σημαντικό ρόλο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πίεση στους δημοσιογράφους, όπως, ε, όπως το παράδειγμα της Σλοβακίας. Και η πίεση αυτή δεν προέρχεται μόνο από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά κυρίως από εσωτερικούς. Οι δημοσιογράφοι πλέον εξαιτία του μειωμένου αριθμού του στα δελτία ειδήσεων πρέπει να παράγουν περισσότερη δουλειά. Επίση, εκφοβισμό. Πολλέ φορέ εκφοβίζονται ή απειλούνται οι δημοσιογράφοι. Ευτυχώ δεν έχουν σημειωθεί ακόμα δολοφονίε δημοσιογράφων. Ευτυχώ το λέω, Έπειτα, τα μέσα ενημέρωσης και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης τους. Ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης, η πολυφωνία, αυτό παίζει σημαντικό ρόλο. Όσο περισσότερα, περισσότερες φωνές ακούγονται, τόσο περισσότερες ειδήσει μπορούν να εμφανιστούν. Μετά, νομικές πτυχές. Η νομοθεσία σχετικά με την ελευθερία έκφρασης, η προστασία των καταγγελτών. η λογοδοσία των μέσων ενημέρωσης είναι επίσης σημαντικό. Μας εμπιστεύεται το κοινό ως δημοσιογράφους πλέον. Ε, και μετά η ελευθερία του τύπου σε γενικές γραμμές. Και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ με αυτό. Η μελέτη εστίασε σε ορισμένες χώρες διότι αυτό μας ζητήθηκε αλλά και το επιθυμήσαμε διότι θέλαμε να δείξουμε την, ε, τις διαφορές ανάμεσα στις ε, διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 27 κρατημέλη έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και οι φωνές είναι διαφορετικές. Ρουμανία. Ας αρχίσουμε με τη Ρουμανία. Με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Στη Ρουμανία πολλοί ερευνητικοί πολλή δουλειά των ερευνητικών δημοσιογράφων γίνεται από ΜΚΟ, διότι πολλές φορές οι δημοσιογράφοι αναγκάζεται να καταφύγουν σε μη κυβερνητικού ε, οργανισμούς για να διεξάγουν το ερευνητικό τους έργο, διότι υπάρχει μεγάλη πίεση, πολιτική πίεση. Να σας φέρω ένα παράδειγμα. Εάν δείτε στο σύνδεσμο Υπήρχε ένα project που έτρεξε από μια μη κυβερνητική οργάνωση επί τέσσερα χρόνια. Στο project αυτό ε, δημοσιογράφοι της περιοχής προσπάθησαν να διερευνήσουν τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην περιφέρειά τους. Οι δημοσιογράφοι λοιπόν αυτοί ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα και αυτό που, ανακάλυψα και αυτό που ανακαλύψαμε και διαπιστώσαμε είναι ότι εάν τους παρέχουμε τα εργαλεία τα κατάλληλα εργαλεία, οι δημοσιογράφοι θα μπορέσουν να φέρουν την είδηση. Αλλά χρειάζονται τη βοήθειά μας, διότι μόνοι τους δεν έχουν τις δυνατότητες να έχουν πρόσβαση ή πολλές φορές δεν ξέρουν πώς να διαχειριστούν τα δεδομένα που έχουν. Μετά στην Ισπανία είχαμε ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική περίπτωση. Η Ισπανία βρίσκεται σε μεγάλη ύφεση και πολύ λίγη προσοχή δίνεται σε οτιδήποτε εκτός της ισπανικής κοινωνίας. Η Ισπανία όμως έχει έναν από τους μεγαλύτερους αλλιευτικούς στόλους παγκοσμίω. Και ένας διεθνής οργανισμός, βασισμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Διεθνές Κονσόρτιο των Ερευνητικών Δημοσιογράφων, και μερικές έρευνες για την αλληλευτική βιομηχανία σε παγκόσμιο επίπεδο και μία από αυτές τις έρευνες αφορούσε τις ε, αλλιευτικές επιχορηγήσεις. Η έρευνα λέγεται «Λαιλατώντας τις θάλασσες». Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η έρευνα αυτή έγινε μόνο επειδή οι Ισπανοί δημοσιογράφοι που ασχολήθηκαν με αυτή την έρευνα είχαν τη βοήθεια των διεθνών αυτών οργανισμών. Και πραγματικά η δουλειά ήταν εξαιρετική και φαίνεται ξεκάθαρα ότι ο αλληλευτικός στόλο δεν χρειάζεται καθόλου επιχορηγήσεις ή τουλάχιστον αυτό που ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούν τις επιχορηγήσεις είναι στην ουσία αποκλειστικά λαιλασία των θαλασσών. Επίσης, κοιτάξαμε τους, ε, την νομοθεσία σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης και πώς αυτό παρεμποδίζει ή βοηθά την ερευνητική δημοσιογραφία. Βρήκαμε ότι παρεμποδίζεται η, δημοσιογραφική, η ερευνητική δημοσιογραφία από την ερευνητικη δημοσιογραφια βρηκαμε οτι παρεμποδιζεται η η ερευνητικη δημοσιογραφια απο την νομοθεσια Όμως η ερευνητική δημοσιογραφία έχει βρει και νέες πλατφόρμες μετάδοσης ειδήσεων. Το διαδίκτυο, για παράδειγμα, στην Ουγγαρία. Η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν διευκολύνει τους δημοσιογράφους στο έργο τους, γιατί πολλές φορές οι εταιρείε που είναι, οι οργανισμοί που είναι αναμεμειγμένοι σε αυτό, τους παρεμποδίζουν. Όμως, τρόπος υπάρχει. Αυτό που ζητούν από εμά οι δημοσιογράφοι της Ουγγαρίας είναι να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα στην, στην Ουγγαρία. Διότι όπως γνωρίζετε ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης δεν βοηθά, δεν εμποδίζει τους δημοσιογράφους, κυρίως όμως δεν τους βοηθά. Έπειτα πήγαμε στο, πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχαμε πληθώρα ειδήσεων. Και όχι μόνο επειδή οι βάσεις δεδομένων είναι στα αγγλικά. Ο τύπος εκεί είναι αρκετά ευρωσκεπτικιστής. Ταυτόχρονα όμως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μία από τις λίγες χώρες όπου υπάρχει μία πολύ μεγάλη βάση δεδομένων. Εκεί είδαμε ότι η συνεργασία μεταξύ δημοσιογράφων πραγματικά είχε αποτελέσματα. Το 2010 έγινε ένα project από το Προεδρείο των Ερευνητικών Δημοσιογράφων, μία μη κυβερνητική οργάνωση, σε συνεργασία με τους ε, Financial Times, το Al Jazeera και το BBC Radio 4. Εξέτασαν πολλές ειδήσει από όλη την Ευρώπη και το project αυτό ονομάστηκε «Τα κρυμμένα εκατομμύρια στην Ευρώπη». Το ρόλο των ε, διαρθρωτικών ταμείων στα κράτη-μέλη και στο σύστημα στο μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαστήκανε έξι μήνες μόνο για να συλλέξουν δεδομένα και να τα κάνουν επεξεργάσιμα. Και θα επανέλθω σε αυτό, ε, περιλαμβάνει μια σύστασή μας, σύσταση στην οποία εσείς μπορείτε να βοηθήσετε. Τα δεδομένα είναι τόσο δυσπρόσιτα, πολλές φορές ε, είναι σε μη επεξεργάσιμες μορφές. Για παράδειγμα, σε PDF, τα οποία είναι κλειδωμένα, τα οποία δεν μπορούμε να ανοίξουμε και να διαβάσουμε. Χρειάστηκαν λοιπόν μήνες για να γίνει αυτή η βάση δεδομένων προσβάσιμη. Προτού αρχίσουμε να εξετάζουμε τα περιεχόμενα της ίδιας της βάσης δεδομένων. Δεν υπήρχαν πάρα πολλά μέσα ή πάρα πολλοί δημοσιογράφοι ε, που είχαν αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους να το εξετάσουν και να αρχίσουν να ζητούν ερωτήσεις. Αυτό λοιπόν που συμπεράναμε είναι ότι χρειαζόμαστε προσβάσιμα δεδομένα και να ασκήσουμε πίεση στις χώρες για να δώσουν τα δεδομένα εγκαίρως ώστε να μπορέσουν οι δημοσιογράφοι μετά να τα επεξεργαστούν. Αυτό το project ήταν αντικείμενο πολύ μεγάλης κριτικής και πολύ δρυμίας κριτικής. Και θέλαμε να το παρουσιάσουμε αυτό με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα, διότι πάντα μπορεί κάποιος να ασκήσει κριτική. Αλλά πρέπει να δούμε και πώς. Εάν κοιτάξετε τους Financial Times, την αναφορά τους στο θέμα αυτό, θα δείτε λεπτομερώς πώς διεξήχθη η έρευνα, θα δείτε τη μεθοδολογία. Και αυτό το project μαζί με τις γεωργικές επιδοτήσεις ήταν το μόνο το οποίο ήταν άριστα διαρθρωμένο. Τώρα πάμε στη Δανία. Η Δανία έχει μία μακρά παράδοση ερευνητικής δημοσιογραφίας, όμως βρήκαμε ελάχιστες αν όχι καθόλου ειδήσει και αναφορές για την απάτη στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και αυτό μας εξέπληξε. Υπάρχει η δομή, όμως Καθώς φαίνεται, οι Δανείοι δεν ενδιαφέρονται για τέτοιες ειδήσει. Και εξεπλάγησαν μάλιστα όταν τους τον αναφέραμε και μας είπαν ότι ναι, καλή ιδέα, θα ασχοληθούμε και με αυτό στο μέλλον. Μετά πάμε στην Ιταλία. Η Ιταλία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πάρα πολλά χρόνια και οι ερευνητικοί δημοσιογράφοι στην Ιταλία διώκονται. Πολλές φορές πρέπει να κρυφτούν αλλά στην Ιταλία πραγματικά κάτι κινείται. Βλέπουμε μικρές πρωτοβουλίες που αναδύονται. Για παράδειγμα, μια πολύ μικρή εφημερίδα, το Φάτο Quotidiano, που άρχισε πριν από δύο χρόνια να εκδίδεται. Υπάρχει, κάτι λοιπόν κινείται και ελπίζουμε να αυξηθούν αυτές οι περιπτώσεις. πολλά, πολλές μάλιστα από αυτές τις μικρές πρωτοβουλίες έχουν και ιστοσελίδα, οπότε είμαστε αισιόδοξοι για την κατάσταση και στην Ιταλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκδίδονται στα αγγλικά. Θα είναι λοιπόν στα αγγλικά, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρει Ιταλικά και δεν μπορεί να το διαβάσει. Βλέπετε λοιπόν ότι διαπιστώνουμε μια μικρή αναγέννηση δημοσιογραφική στην Ιταλία η οποία εξαπλώνεται σιγά σιγά στην Ευρώπη. Και μπορούμε να δούμε και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σε ορισμένα θεσμικά όργανα διαπιστώνεται μεγάλη επιθυμία για συνεργασία με την ερευνητική δημοσιογραφία, το δίκτυο επικοινωνίας της Όλαφ, το οποίο ξεκίνησε το 2004 για παράδειγμα. Είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα. Είδαμε ότι πολλοί δημοσιογράφοι εκτιμούν ιδιαίτερως αυτή την πρωτοβουλία και μπορεί αυτή να θεωρείται μια, και να θεωρηθεί ως μια βέλτιστη πρακτική και για τους υπόλοιπους εργαζόμενοι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πράγματι προσπαθούν να συνεργαστούν και όταν η Όλαφ ε, διενεργεί έρευνες ε, επί διαφόρων προγραμμάτων και σχεδίων και δαπανών ε, κοινοτικού χρήματος είναι δύσκολο να πει από πού άτλησε τις πληροφορίες και τα στοιχεία που έχει. Δεν μπορεί να το πει από τη στιγμή που συνεχίζουν να διενεργούνται τέτοιου είδους έρευνες και τελικά χρειάζεται πάρα πολλής χρόνο στα κράτη-μέλη μέχρι ότου καταλήξουν σε κάποιο οριστικό συμπέρασμα. Παρόλα τα αυτά διαπιστώνεται μεγάλη όθηση, επιθυμία ε, να ε, κινηθούν τα πράγματα ε, προς τα εμπρός μεταξύ υπαλλήλων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και δημοσιογράφων, ερευνητών δημοσιογράφων. Δεν θα πω ότι είναι οι καλύτεροι φίλοι, αλλά είναι σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η κινητικότητα. Θα ήθελα τώρα να ε, πω τα βήματα που να μιλήσω για τα βήματα που θα πρέπει, να, θα πρέπει να γίνουν. Λένε οι δημοσιογράφοι ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Αυτό ε, δεν είναι δικαιολογία. Είναι θέμα προτεραιοτήτων και οργάνωσης. Μην δεχτείτε ε, αυτή την απάντηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν είχαμε παραπάνω χρήματα αυτό δεν θα μας βοηθούσε. Και βέβαια θα μας βοηθούσε. Πολύ συχνά διαπιστώσαμε διστακτικότητα από πλευρά ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Έλεγαν δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα σε δημοσιογράφους. Όχι, η αλήθεια είναι ότι μπορείτε να δώσετε χρήματα σε δημοσιογράφους τη στιγμή που μπορείτε να δείξετε ότι δεν υπάρχει σύνδεση με τα θέματα που θα καλύψουν και χρειάζονται τη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Αυτό πράγματι ε, θα έχει μεγάλη διαφορά στα θέματα που καλύπτει η ευρωπαϊκή δημοσιογραφία. Μπορείτε να εξετάσετε τέτοιου είδου πρωτοβουλίες και πράγματι αξίζει αυτό και θα παρουσιάσουμε ε, και τέτοιου είδους επιχειρήματα. Λοιπόν, ε, σιγά σιγά αλλάζει το ραντάρ της ευρωπαϊκής δημοσιογραφίας και αρχίζει και εντοπίζει περισσότερο τα σήματα της Ευρώπης. Ε, λόγω της κρίσης δεν μπορεί κανείς δημοσιογράφος να πει ότι το, η Ευρώπη σαν θέμα δεν είναι ενδιαφέρον, δεν είναι ψηλά στις προτιμήσεις των τηλεθεατών ή των αναγνωστών. Οργανώσαμε μία διάσκεψη, ένα συνέδριο προ ολίγου καιρού με τίτλο «Από πότε η εξουσία συνεδριο προ λιγου καιρου με τιτλο βαρετή» Ακριβώς για να καταπολεμήσουμε αυτό το στερεότυπο ότι τα της Ευρώπης, το ευρωπαϊκό γίγνεσθε είναι τόσο βαρετά σε σχέση με τον Ευρωπαίο πολίτη. Κανείς λοιπόν δεν μπορεί πια να το ισχυρίζεται αυτό ε, λόγω της κρίσης. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε να επιμένουμε ώστε τα θέματα που καλύπτουν την ευρωπαϊκή δυσιογραφία να συνεχίσουν να είναι υψηλής προτεραιότητας ε, στα ε, γραφεία σύνταξη των δημοσιογράφων. Γιατί πράγματι ε, θέλει ο Ευρωπαίος πολίτης να ξέρει πώς ξοδεύεται το, το χρήμα που πληρώνει, το ευρωπαϊκό χρήμα και γι' αυτό πρέπει συνεχώς να πιέζουμε ε, τους δημοσιογράφους να μην στρέφουν την προσοχή τους μακριά από τα ευρωπαϊκά θέματα. Πάρα πολλά χρήματα ευρωπαϊκά στρέφονται προς την κατάρτιση και εκπαίδευση των δημοσιογράφων. Αυτό πρέπει να το δείτε, πρέπει να το ερευνήσετε. Για πού ξοδεύονται αυτά τα χρήματα. Πολύ συχνά τα προγράμματα, οι σχέδια είναι ανόητα και δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι δημοσιογράφοι. Μιλήστε με τους δημοσιογράφους που χρειάζονται εκπαίδευση και ρωτήστε τους τι πραγματικά χρειάζονται. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα μπορούν να βοηθήσουν εμάς τους δημοσιογράφους και εμείς μπορούμε να βοηθήσετε εσάς, να βοηθήσουμε εσάς ε, στην διατήρηση στοιχείων, στην, στους φακέλους, στην τήρηση φακέλων και συστημάτων για το πώς δαπανώνται αυτά τα κονδύλια. Και η μη συμμόρφωση με ε, ε, με τα πεπραγμένα και με αυτά που πρέπει σε ευρωπαϊκό θεσμικό επίπεδο μπορεί να τιμωρείται. μπορείτε να μας βοηθήσετε και στο εξής. Να επιταχύνουμε ε, τη διαδικασία πρόσβασης σε έγγραφα ε, και ε, σε πηγές. Προστασία της πηγής, των πηγών μας, σφύριγμα της φυρίχτρας. Όλα αυτά γίνονται με άνισο τρόπο στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να υπάρχει μια εξίσωση. Γραπτός τύπος και πλουραλισμός. Η, Επίτρο... Επίτροπος Κρούζ κάνει πολλά για αυτό το θέμα και τη στηρίζουμε γιατί ο πλουραλισμός στα μέσα μαζικής επικοινωνίας είναι εξαιρετικά σημαντικός. Εάν έχετε μόνο μη έναν ή δύο ε, μεγιστάνες που συγκεντρώνουν όλες τις εφημερίδες και ε, τον τύπο και μετά αυτοί δεν θέλουν να δημοσιεύσουν τη χύψη ιστορία, το χύψη θέμα, υπάρχει πρόβλημα. Όσο περισσότεροι λοιπόν τόσο καλύτεροι εθνική δημόσια τηλεόραση, εθνικό δημόσιο ραδιόφωνο, εμπορική ιδιωτική τηλεόραση, ε, κανάλια εκπομπής και ειδησιογραφίας και τύπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σε, όλους, όλα αυτά τα πεδία μπορεί η ερευνητική δημοσιογραφία να ενισχυθεί και να ανθίσει. Και έχουμε και τη δουλειά με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που εργάζονται και συνεργάζονται με δημοσιογράφους ώστε να προβληθούν αυτά τα ευρωπαϊκά θέματα. Είναι πολύ σημαντικό όλα αυτά και αν δουλέψουμε μαζί θα καταφέρουμε οι ειδήσει αυτές να προβληθούν. Συμπερασματικά, έξι μήνες δουλειάς στην ερευνητική δημοσιογραφία με διδάσκουν το εξή. Να δοθεί προτεραιότητα, να υπάρξει αποφασιστικότητα και να υπάρξει συνεργασία. Αυτές είναι οι τρει λέξεις κλειδιά ώστε η ερευνητική δημοσιογραφία πράγματι να συμβάλλει στο να αποτραπεί η απάτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να είναι λιγότερο ε, δύσκολο να πιστούν οι συντάκτες, οι διευθυντές των ειδήσεων για το την ανάγκη να συμπεριληφθεί το ε, χύψη θέμα στην ε, η δημοσιογραφία Θα πρέπει να δίδεται περισσότερη προτεραιότητα στα ευρωπαϊκά θέματα ως προς την κάλυψη τη δημοσιογραφική. Θα πρέπει όλοι να προσέχουμε και να ενδιαφερόμαστε περισσότερο για όλα αυτά τα θέματα. Και όσοι ε, εργαζόμενοι ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πρέπει να απαντούν σε δημοσιογράφους που ρωτούν για το πώς δαπανώνται συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κονδύλια, πρέπει να είναι πιο επιμελής και να μεριμνούν να απαντούν εγκαίρως και με ακρίβεια. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να κάνουν περισσότερα. Δεν θα πρέπει να αποφεύγουν τις ερωτήσεις και να παραπέμπουν στο χύψη ε, έγγραφο ή οτιδήποτε, γιατί δεν, θέλουμε, δεν θέλουμε να, αφήθ, να αφαιθεί χώρο στους δημοσιογράφους να ε, βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Εάν είστε ακριβεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τότε το θέμα θα καλυφθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια από τον εκάστοτε δημοσιογράφο. Και Πρέπει να αναπτύξουμε συγκεκριμένες δεξιότητες των ε, ερευνητών δημοσιογράφων, οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να δραστηριοποιηθούν σε αυτό το τομέα. Άλλωστε, θα είναι πιο εύκολο να καλυφθούν όλα αυτά τα θέματα όταν θα υπάρξουν περισσότερες διαθέσιμες πηγές, έγγραφα και υλικό τεκμηρίωσης γενικότερα. Οι δημοσιογράφοι θεωρούν ότι πράγματι η στενή συνεργασία βοηθάει. Ε, ανέφερα το ισπανικό παράδειγμα και το βρετανικό παράδειγμα. Βοηθάει η συνεργασία. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε. Πρέπει ε, να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Το ξέρω ότι οι δημοσιογράφοι κυνηγούν πάντοτε το λαβράκι, το δημοσιογραφικό λαβράκι. Όμως πρέπει να συνεργαστούμε μεταξύ μας και με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και ε, με τον τύπο. Εάν επιτευχθεί ομοιομορφία στην ε, ε, αναφορά των στοιχείων στα κράτη-μέλη, τότε θα ε, γλιτώσουμε πάρα πολύ χρόνο. Η δουλειά ερευνητική του δημοσιογράφου θα γίνεται πολύ πιο γρήγορη και δεν θα γίνονται και τόσα λάθη και δεν θα χρονοτριβούν τόσο πολύ οι δημοσιογράφοι, πράγμα για το οποίο κατηγορούνται πολύ συχνά. Αν υπάρχει δηλαδή μια ομοιόμορφη αναφορά από πλευρά κρατών μελών, αυτά θα τα επεξεργάζονται και θα τα παρουσιάζονται καλύτερα οι δημοσιογράφοι. Άλλωστε, ο υπέρτατος δικαιούχος αυτού του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου είναι ο Ευρωπαίος πολίτης. Βεβαίως όλα αυτά τα βήματα δεν μπορούν να είναι τα ίδια για όλους. Δεν είναι ένα μέγεθος ε, κουστούμι που μπορεί να το φορέσει οποιοδήποτε. Κάποια χρειάζονται στους μεν και κάποια άλλα βήματα χρειάζονται στους δε. Είναι όμως σημαντικά ώστε να εδρεωθεί εμπιστοσύνη, σεβασμός μεταξύ ε, δημοσιογράφων και ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ούτως ώστε ούτε οι τελευταίοι να αποφεύγουν να απαντούν, ούτε οι πρώτοι δημοσιογράφοι να ερμηνεύουν τις απαντήσεις κατά το δικό τους δοκούν. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω σε αυτό το Σολυμίο την Επιτροπή σας για την ευκαιρία που μου έδωσε να διεξάγω όλη αυτή την ερευνητική δραστηριότητα και με χαρά θα απαντήσω σε όσες ερωτήσεις τυχόν έχετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σμιτ. Πραγματικά εκτενέστατη η παρουσία σας, η εισήγησή σας. Ε, βλέπω ότι οι συναδελφοί ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτά που είπατε. Ήδη εννέα έχουν ζητήσει το λόγο. Αυτό και μόνο λοιπόν το γεγονός αποδεικνύει ότι ε, θέσατε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Αλλά σας παρακαλώ όλοι οι ερωτώντες ε, να υποβάλουν συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σμιτ και αγαπητοί συνάδελφοι δεν θέλω σε καμία περίπτωση να στερήσω από τους συναδέλφους μου ε, τη δυνατότητα να πάρουν το λόγο, ε, μας λέει ο κύριος Ντόιτς. Θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένος, να κάνω ένα σχόλιο και ενδεχομένως να θέσω δύο-τρία ερωτήματα. Πρώτον, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον διάβασα τη μελέτη σας, την έρευνά σας. Αυτό σας το επιβεβαιώνω. Και από τη στιγμή που οι συγγραφείς είναι παρόντες, ε, θέλω να δηλώσω ξεκάθαρα ότι απογοητεύτηκα πλήρως. Και το επαναλαμβάνω αυτό. Απογοητεύτηκα πλήρως. Είμαι τρία χρόνια βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρώτη φορά βλέπω να παρουσιάζεται μελέτη έρευνα σε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία να σέβεται τόσο λίγο να τη ε, ακολουθεί τόσο λίγο, τόσο ελάχιστα ε, ε, τα επαγγελματικά επίπεδα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ επιφανειακή. Δεν διατυπώνεται καμία πρόταση, δεν διατυπώνεται καμία σύσταση. δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι καινοτόμο, τίποτα το οποίο να είναι καινούριο για το θέμα της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Τίποτα δεν μαθαίνουμε που δεν ξέραμε ήδη. Είτε οριζόντια είτε κάθετα. Ε, είναι μία συλλογή γενικοτήτων, ε, γενικεύσεων, Είναι μία βάση δεδομένων από 233 άρθρα. Πώς μπορείτε μία συλλογή 233 άρθρων να την αποκαλείτε βάση δεδομένων. Στην Ουγγαρία έχουμε 6-7 άρθρα. Δηλαδή μιλούμε για δημοσιογράφους τους οποίους εσείς έχετε ε, ε, ερωτήσει Άρα καταλαβαίνω ότι είναι οι δημοσιογράφοι που ήθελαν να είναι παρόντες μόνο και να στερήσουν από τους άλλους δημοσιογράφους ε, αυτή τη δυνατότητα. Να πούν και αυτή τη γνώμη τους. Στην Ουγγαρία τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των άρθρων για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων έχει ξεπεράσει ε, το 100 πάνω από 100 άρθρα λοιπόν. Εμπλήρη πλήρη γνώση αυτών των αριθμητικών στοιχείων μπορώ να πω ότι δεν είναι σοβαρό ενώ υπάρχουν πάνω από 100 να δουλεύετε με 6, πάνω σε 6-7 άρθρα μόνο. Και επίσης δεν έχετε ασχοληθεί καθόλου στη μελέτη σας, στην έρευνά σας με την προσβασιμότητα, την προσβασιμότητα στα δεδομένα. Ε, στα κράτη-μέλη. Μόνο τους δημοσιογράφους ρωτήσατε. Δηλαδή, είναι σαν να είχατε ρωτήσει μόνο τους γιατρούς αν, θέλατε να κάνετε έρευνα για το εκάστοτε Εθνικό Σύστημα Υγείας, χωρίς να μιλήσετε και στους άλλους χρήστες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Από εκεί και πέρα. Ε, δεν μάθατε ποτέ αν υπήρξαν ε, ε, διοικητικές διώξεις, αν τελικά βγήκαν πορίσματα στην Ουγγαρία, για την Ουγγαρία αναφέρεται τον ε, νόμο για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Είναι εξαιρετικά της μόδας να βγαίνει ο καθένας και να επικρίνει αυτό ε, το νόμο ε, περί μέσων μαζικής επικοινωνίας στην ε, Ουγγαρία. Γιατί όμως δεν αναφέρεται και τους δύο κανόνες οι οποίοι είναι πρότυπο στην Ευρώπη, ότι δηλαδή δεν μπορεί η δικαιοσύνη να ασκήσει καμία δίωξη σε καμία περίπτωση στον ερευνόντα δημοσιογράφο ε, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, κανόνες που είναι πραγματικά εχέγγυα ε, για τη δημοσιογραφία ε, και δεν υπάρχουν σε κανένα άλλο κράτος. Και μάλιστα ε, υπάρχει και κανόνας που λέει ότι αν ο δημοσιογράφος δεν σέβεται, δεν τηρεί τον νόμο, όταν αποκτά συγκεκριμένη πληροφορία, αν τελικά αποδειχθεί ότι η πληροφορία ήταν χρήσιμη για το κοινό, ήταν προ όφελο του κοινού αγαθού, του κοινού ωφέλου, τότε δεν μπορεί να διωχθεί ο δημοσιογράφο για την αθέμητη ή παράνομη πρόσβαση στην πληροφορία, αφού τελικά αυτή αποδείχθηκε υποφελή. Αυτά λοιπόν είναι κανόνε που είναι πραγματικά εχέγγυο ε, για τη δουλειά του δημοσιογράφου και δεν του αναφέρεται καθόλου. Λυπούμε ε, ε, λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, για το περιεχόμενο της έκθεσής σας, ειδικά σε ό,τι αφορά την Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, ακούσαμε ακούσαμε τον πρώτο μιλητή, ο κύριος Ετσενίκη. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εσείς είπατε ότι εμφανιστήκατε με δύο ιδιότητες ως πρόεδρος της Επιτροπής και ως εισηγητής. Ε, και εγώ έχω δύο ιδιότητες, ε, την πολιτική ιδιότητα και τη δημοσιογραφική. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η συζήτηση είναι καθοριστική σημασίας έγινε λόγος, αναφέρθηκε το θέμα της σημερινής εποχής. Ε, υπόθηκε ότι πάρα πολλοί δημοσιογράφοι δεν αναφέρονται στα σκάνδαλα και κυρίως αυτά που έχουν σχέση με την ε, κατάχρηση των κοντιλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί αν το κάνουν αυτό, αυτό θα εκλειφθεί ως ε, δυσφήμιση της δικής τους της χώρας. Αυτό συμβαίνει και στη δική μου τη χώρα, την Πολωνία. Ε, υπάρχει συνεχής ε, δυσφήμιση της ε, χώρας μας. Ε, πολλές φορές αναφέρεται ότι η Πολωνία καταχράται αυτών των κοντιλίων. Δεν είναι αλήθεια. Ε, δεν είναι αλήθεια αυτό καθόλου. Εμεί χρησιμοποιούμε σωστά τα κονδύλια και ε, ο λόγο όμως όλου αυτού του περιγύρου είναι πολύ δύσκολο ε, να ενισχυθεί η ερευνητική δημοσιογραφία. Πριν από κάποιε ημέρε έγινε κάποιο τεστ για να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι γνωστά τα κονδύλια που χορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από νέα λοιπόν χρόνια, τότε ε, αναφέρεται ότι θα έπρεπε να λέγονται μόνο καλά λόγια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε υπήρχε αυτή η γραμμή, δηλαδή ότι έπρεπε να αναφέρονται μόνο τα ε, υπέρ και ποτέ τα μειονεκτήματα, τα κατά της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εσείς λοιπόν μιλήσατε και για αυτή την συμβίωση που προκύπτει ανάμεσα στους ε, δημοσιογράφους και τους ε, αξιωματούχους. Τα πράγματα όμως είναι λιγάκι διαφορετικά, δεν είναι έτσι ακριβώς. Οι αξιωματούχοι είναι εκείνοι που πολλές φορές ε, προκαλούν σκάνδαλα και δεν αναφέρομαι σε αυτούς των Βρυξελών, αλλά αναφέρομαι κυρίως σε αξιωματούχους εθνικού και τοπικού επίπεδου στα κράτη-μέλη. Πρόσφατα στην Πολωνία δημοσιεύτηκαν άρθρα που αφορούν σε μια ολόκληρη σειρά περιπτώσεων όπου υπάλληλοι της ε, τοπικής αυτοδιοίκησης ε, οι οποίοι λαμβάνουν κονδύλια της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης καταχρώνται αυτά τα χρήματα τα μοιράζουν μεταξύ τους, ε, στους συγγενείς τους. Ε, νεποτισμός λοιπόν ε, σε όλη του την μεγαλοπρέπεια. Και έχει γίνει λόγος για περιπτώσεις όπου οι πάλι αυτή της τοπικής αυτοδίκης έχουν προσλάβει τη σύζυγό τους ή κάποιο άλλο συγγενικό τους πρόσωπο ως συνεργάτη. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι περιπτώσεις. Εγώ τώρα δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά θέλω να πω το εξής. Ένας δημοσιογράφος στη δική μου τη χώρα, καθότι οι αξιωματούχοι και οι πολιτικοί προάγουν νόμους οι οποίοι κατάφορα παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία. Είχαμε στην αρχή το πρόβλημα του αυτοκινητόδρομου ε, κατόπιν το πρωτάθλημα του 2012. Εδώ μάλιστα ε, μας επισκέφθηκε και ο πρώην Υπουργός. Ε, εδώ υπάρχει και ο κύριος Λιμπεράτσκι. Ο κύριος Λιμπεράτσκι είναι πρώην Υπουργός στη χώρα μου. Ίσως μπορεί να τοποθετηθεί από αυτού που λέω. Τι έγινε λοιπόν σχετικά με το σκάνδαλο αυτό. Τελικά το κράτος αποζημίωσε τις επιχειρήσεις και αυτό προφανώς είναι παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιληφθεί του θέματος αυτού. Αυτά που είπε ο συνάδελφος κύριος Ντότσε, ίσως ε, να έχει δίκιο όσον αφορά σε κάποιες ε, πτυχές της ε, έκθεσης αλλά το να μιλάει κανείς ε, για την ε, ερευνητική δημοσιογραφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή η μορφή δημοσιογραφίας είναι απολύτως απαραίτητη ακόμα και αν μερικές φορές αυτή η μορφή δημοσιογραφίας έρχεται σε σύγκρουση με εθνικές ε, εκστρατείες που δεν θέλουν να αποκαλύπτονται σκάνδαλα για να μην δυσφημείται η χώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κοιτάξτε, ο κύριος Λιμπεράτσκι έχει το λόγο. Είχε ζητήσει το λόγο έτσι κι αλλιώς. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω πολωνικά. Κοιτάξτε, σήμερα συζητάμε για το θέμα αυτό και έχω να σας ε, κάνω μία ερώτηση προς ε, τους συντάκτες της ε, έκθεσης. Καταρχήν, υπάρχει ευρέως αποδεκτός ορισμός του, ε, της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Και εάν υπάρχει τέτοιου είδους ε, ορισμός, ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτού, αυτής της μορφής δημοσιογραφίας και της δημοσιογραφίας γενικότερα. Και επίση, θέλω να ρωτήσω, όταν ε, λέει ένας δημοσιογράφος, εγώ ασχολούμαι με την ερευνητική δημοσιογραφία τι ακριβώς εννοεί. Γιατί εδώ δείτε ένα πολύ βασικό θέμα. Ε, είναι το θέμα της ευθύνης που ανέφερε και ο κύριος Ντόιτς. Ε, είναι πολύ σημαντικό να λειτουργεί κανείς υπεύθυνα, να μην φοβάται τα γεγονότα, να μην φοβάται την τιμωρία, διότι ενδέχεται να αποκαλύψει κάποια στοιχεία. Απ' την άλλη φορά βέβαια ε, δεν πρέπει να δέχεται να τον καπελώνουν όπως λέμε απλά, να μην δέχεται να ε, γίνεται παιχνίδι στα χέρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης και της ε, κυβέρνησης. Ε, σε διάφορα κράτη-μέλη έχουμε κάνει εμπειρία, πολλές εμπειρίες. Ο συνάδελφός μου αναφέρθηκε στην Πολωνία, δεν αναφέρθηκατε εσείς, αλλά το είπε ο συνάδελφος. Πάντως, όχι μόνο στην Πολωνία, αλλά παντού είναι απαραίτητο να υπάρχει η ερευνητική δημοσιογραφία. Και όσον αφορά τα συμπεράσματά σας, τελικά τι γίνεται ακριβώς με τα κοινοτικά κονδύλια. Ε, κάπου γίνεται αναφορά στην έκθεσή σας ότι πολλές κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τα κοινοτικά κονδύλια κατά κύριο λόγο για να ε, αποκτήσουν φιλίες ε, με εταιρείες ε, δημοσίων σχέσεων και αυτό ισχύει κατά κύριο λόγο στην Πολωνία. Το Υπουργείο Γεωργίας προάγει ένα πρόγραμμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και προσπαθεί να πείσει την κοινωνία ότι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσφέρει όλες τις απαντήσεις και θα λύσει τα προβλήματα των γεωργών. και επίσης ε, προσπαθούν να πείσουν ότι ε, πρέπει να ε, προωθηθεί η κοινωτική νομοθεσία έτσι ώστε να είναι όλοι ευχαριστημένοι στην πολωνική κοινωνία. Το θέμα που τίθεται είναι πού μπαίνουν τα όρια και σε ποιο βαθμό η ερευνητική δημοσιογραφία είναι πραγματικά υπεύθυνη. Πότε θα πρέπει να την χάνει προστασίας, αλλά την ίδια στιγμή η δημοσιογραφία αυτή να μην είναι ανεύθυνη. Η διαφορά ανάμεσα αυτά τα δύο είναι πολύ λεπτή. Μερικές φορές καλές οι προθέσεις, αλλά δεν ε, είναι πάντα το καλύτερο. Είναι θέμα λοιπόν καλής βούλησης και ισορροπίας ε, μεταξύ ευθύνη και εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το γεγονός ότι συζητάμε σήμερα αυτό το θέμα. Πρέπει να αποδείξουμε ότι τα κοινωτικά κονδύλια ε, εκταμιεύονται με διαφανείς κανόνες. Ποιος τα παίρνει, γιατί, πώς, πώς τα διαχειρίζονται αυτοί που τα εισπράττουν. Πολύ συχνά λοιπόν ακούω ότι πρέπει να ε, εκταμιεύουμε τα κοινοτικά κονδύλια, ε, να τα εντάσσουμε στις δαπάνες. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Όχι, τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μην εντάσσονται στις δαπάνες, αλλά στις επενδύσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρώ ότι όταν μιλάμε για ερευνητική δημοσιογραφία θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον ε, συνάδελφο που με αντικατέστησε. Ε, τώρα λοιπόν θα συνεχίσουμε με τους επόμενους ομιλητές. Και επειδή περνάει η ώρα, θα ήθελα παρακαλώ ε, να μην ξεχνάτε το ρολόι. Και η συνάδελφος Βενίνη, από ο συνάδελφος, με συγχωρείτε, ο συνάδελφος, η συνάδελφος Σαρχεντίνη είναι από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Ευχαριστώ. Άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τα λόγια της κυρίας Σμιτ και άκουσα και με πολύ μεγάλη προσοχή τους συναδέλφους μου. Πρέπει να γνωρίζουμε το εξής. Μια δημοκρατία που λειτουργεί πρέπει πράγματι να μεριμνά ώστε να υπάρχει και αντίλογος. Να μπορούν να ακουστούν οι φωνές που διαφωνούν να υπάρχει πολιτικός έλεγχος. Και ε, αυτοί που ελέγχουν πρέπει και αυτοί να ελέγχονται. Ούτως ώστε να υπάρχει προστασία. και να μπορούν να υπάρχουν άρθρα επικριτικά ή συγκαταβατικά για το γίγνεσθε στις Βρυξέλλες. Άκουσα συναδέλφους να λένε ότι η έρευνα δεν περιλαμβάνει τίποτα το καινούριο. Όμως, πρέπει να διευκολύνουμε τις δραστηριότητες των δημοσιογράφων που ασκούν ερευνητική δημοσιογραφία και πρέπει να διαβεβαιωθούμε να βεβαιωθούμε ότι ε, έχουμε πλουραλισμό στα μίντια πολλά μίντια σε κάθε χώρα. Κάθε χώρα έχει τις δικές της συνήθειες, κάθε δημοσιογραφία έχει τις δικές της συνήθειες σε κάθε χώρα. Ο πλουραλισμός είναι το πιο σημαντικό. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την κυρία Ρέντιν να προτείνει μια οδηγία για το πλουραλισμό στα μίντια. Μπορεί αυτό να μην έγινε, όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε νομοθεσία ώστε να προστατεύεται η ποικιλότητα, η διαφοροποίηση των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Κάθε φορά μας λένε ότι αυτό θα ήταν εξαιρετικά δαπανηρό, αλλά εγώ συνεχίζω να μην καταλαβαίνω γιατί θα ήταν τόσο πια δαπανηρό, υποτίθεται. Θα πρέπει επίσης να δεχόμαστε τους ελέγχους. Στην ανάλυση σας, κάτι το οποίο θεωρώ εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το εξής. Μεταξύ των 27 κρατών μελών με διαφορετικό τρόπο γίνεται η διαχείριση της πρόσβασης στα, έγγραφα, γίνεται ο έλεγχος ε, της δημόσιας εξουσίας. Είχαμε την ευκαιρία εδώ να συζητήσουμε τον τρόπο πρόσβαση στα έγγραφα του Συμβουλίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάναμε πάρα πολλά. Είδαμε ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενδεχομένως χρονοτριβούσαν, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε καταλήξει σε ένα status quo σε μια καθεστική κατάσταση. Επομένως, ενδεχομένως υπάρχει άλλος τρόπος, ε, ένας τρόπος να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, ώστε να έχουν οι δημοσιογράφοι πρόσβαση σε ποιοτικά στοιχεία, σε ποιοτικέ πληροφορίες, ώστε να αλλάξουν οι νοοτροπίες και εδώ στις Βρυξέλλες και ε, στις πρωτεύουσες από πλευράς δημοσιογράφων. Είναι δύσκολο και δεν έχει νόημα να λέμε ότι εμείς θα κάνουμε αυτό που κάνουμε και εσείς να βρείτε τρόπο να μπείτε ή να αποκτήσετε πρόσβαση. Ευχαριστώ, κύριος Βόγκαν. Ευχαριστώ. πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ερευνητέ για την δουλειά που έκαναν. Η συζήτηση ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, είναι διαφορετική από αυτό που συζητούμε συνήθως αυτήν εδώ την Επιτροπή. Γι' αυτό και ενδιαφέρει τόσο πολύ τους συναδέλφους το θέμα. Θα ήθελα να σας δώσω τη δική μου άποψη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Νομίζω πως όλοι θα συμφωνήσουν ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ελεύθερο τύπο. Ελεύθερο και ανεξάρτητο επίσης τύπο. Νομίζω πως κανείς δεν θα μπορούσε να πει τον βρετανικό τύπο ανεξάρτητο. Όχι. Ανήκει σε ορισμένου εύπορου ανθρώπου, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν μένουν καν εκεί και οι περισσότεροι δεν είναι απλά δεξιοί, αλλά αρκετά δεξιοί και πολλοί ευρωσκεπτικιστές. Γι' αυτό ε, βλέπουμε πολλές ε, ειδήσει, πολλά άρθρα στο Βρετανικό τύπο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι οι δημοσιογράφοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα όχι επειδή θέλουν να βοηθήσουν, όχι επειδή θέλουν να είναι δημοκρατικοί, αλλά επειδή θέλουν να ασκήσουν κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτό που εμείς εδώ κάνουμε σε πολλά άρθρα καθημερινά ε, διαφαίνεται αυτό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. ω εισηγητής για τον ε, προπολογισμό του Κοινοβουλίου στην ε, τελευταία ολομελία μίλησα ε, για αυτό και μετά από μια ψηφοφορία η επικεφαλίδα στις εφημερίδες ήταν οι ευρωβουλευτές ψήφισαν για τον εαυτό τους μια τεράστια παχυλή αύξηση. Κανείς δεν ψήφισε τέτοια αύξηση. Η αύξησή μας μαζί με τις αυξήσεις των υπόλοιπων υπαλλήλων αποφασίζεται και εγκρίνεται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Τίποτα δεν υπήρχε στην έκθεση που ψηφίστηκε για το μισθό, για το ότι εμείς αυξήσαμε τον ίδιο, τις ίδιες μας τις αποδοχές. Και να πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο διεξάγεται μια δικαστική έρευνα σχετικά με τον ρόλο του τύπου μετά από τα πρόσφατα σκάνδαλα όπου οι δημοσιογράφοι παραβίασαν άρδιν την, ε, την ιδιωτική ζωή των ανθρώπων και σε πολλές φορές κατέστρεψαν ζωές. διότι αυτό που θέλουν είναι να πουλήσουν φύλλα και, αυτό, και γράφουν ιστορίες για να πουλήσουν, που πολλές φορές δεν είναι αληθινές και πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορώ να τους αποκαλέσω όλους δημοσιογράφους, ε, δυστυχώς υπάρχουν και πρέπει να τους λάβουμε υπόψη. Έχω και γι' αυτό μια ερώτηση για τους ε, μελετητές. Θα μπορέσετε να λάβετε υπόψη σας αυτές τις πολιτικές ε, πτυχές, θα μπορέσετε να λάβετε υπόψη τις απόψεις των δημοσιογράφων με τους οποίους μιλήσατε στο Ηνωμένο Βασίλειο, διότι φυσικά πρέπει να εξετάσουμε και το background και το συγκείμενο. Ευχαριστώ πολύ επόμενος είναι ο κύριος Έρενχάουζα και μετά ακολουθούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Κύριε Ερενχάουζα, ευχαριστώ πολύ. Σύντομος και περιεκτικός θα είμαι. Στην μελέτη αναφέρεστε σε έναν αριθμό 80 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην, έρευνα της, στην ερευνητική δημοσιογραφία. Να αναφέρω ότι το 2% διοχετεύτηκε. Εγώ θέλω να ρωτήσω ότι αυξήθηκε κατά 2%. Εγώ θέλω να ρωτήσω πώς έγινε αυτό, πώς μπορούμε αυτά τα 80 ε, εκατομμύρια δολάρια να τα ανακατανέμουμε για την καλύτερη λειτουργία της ε, ερευνητικής δημοσιογραφίας και των προγραμμάτων. Επίσης, όσον αφορά τη διαφάνεια, πώς θα πώς εμείς διαθέτουμε τα δεδομένα στη διάθεση των δημοσιογράφων, με ποια μορφή. Και επίσης, σε ποιους πολυστομητικείς ε, είδατε, διακρίνατε εσείς θετικά στοιχεία και η Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται, σε ποιο σημείο βρίσκεται όσον αφορά τη διάθεση δεδομένων και σε σχέση με τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μούλνα την... έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα υπόθηκαν. Θα είμαι λοιπόν σύντομος. Δύο ερωτήσεις. Καταρχάς αναφέρατε τους καταγγέλτες. Πόσο σημαντική είναι αυτή. Και υπάρχει νομοθεσία που, που αρκεί για να τους προστατεύσει. Έπειτα, μια διαφορετική κάπως ερώτηση οι ίδιοι οι δημοσιογράφοι εποφελούνται, απολαμβάνουν αρκετής προστασίας από την νομοθεσία στα διάφορα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μούλτερ. Επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση και για την παρουσίαση. Η συζήτηση αυτή μου φαίνεται σαν το τρίγωνο των Βερμούδων κάπως. Φυσικά το τρίγωνο έχει τρεις πλευρές. Τους πολιτικούς, τον τύπο και το κοινό. Οι πολιτικοί τα έχουν βάλει με τον τύπο γιατί δεν γράφει αρκετά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέσα λένε πως δεν έχουν αρκετά άρθρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν ενδιαφέρει το κοινό, το αναγνωστικό κοινό. Και το κοινό λέει ότι δεν ενδιαφέρεται για την Ευρωπαϊκή Ένωση διότι δεν γνωρίζει αρκετά ούτε από τους πολιτικούς ούτε από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι ένα μπούσουλο για το πώς θα βγούμε από αυτό το τρίγωνο των Βερμούδων και, το, και να προσπαθήσουμε να ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον του κοινού για την Ευρωπαϊκή Ένωση, για, αυτά που κάνουμε εδώ. Ήταν εξαιρετική παρουσίαση των στατιστικών. Το ερώτημα όμως που έχω είναι, είναι εάν αυτό αρκεί ή εάν πρέπει να κοιτάξουμε ευρύτερα το θέμα, να δούμε το συγκείμενο. Α παραδεχτούμε ότι η δομή της Ευρωπαϊκής Ένωση είναι αρκετά περίπλοκη. Η συνθήκη της Λισαβόνα, για παράδειγμα, είναι ευανάγνωστο έγγραφο. Είναι. Αλλά η διαδικασία λήψη αποφάσεων είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Είναι πολύ δύσκολο να να μάθει κανεί πώ λαμβάνονται οι αποφάσει και όχι μόνο για του δημοσιογράφους αλλά και για το κοινό. Και αυτό δυσχεραίνει την, ε, το, την ανάπτυξη ενδιαφέροντος στο κοινό. Ας δούμε λοιπόν το ευρύτερο πλαίσιο του πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Και τώρα η δεύτερη, μας είπατε, δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει χρήμα, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν λόγια, δεν γράφεται τίποτα. Ναι, δεν υπάρχουν επιχειρήματα. Θα έπρεπε όμως να υπάρξουν επιχειρήματα. μπορείτε για παράδειγμα, ναι, μπορείτε στον ελεύθερο χρόνο σας να ασχολείστε με την ερευνητική δημοσιογραφία. Αν δείτε όμως τις εφημερίδες τις, κύρι, τις ε, μεγάλες εφημερίδες, θα δείτε ότι είναι επιχείρηση και ως κάθε επιχείρηση τους ενδιαφέρει το κέρδος, η δημοσιότητα. Το κέρδος προκύπτει από τη δημοσιότητα, οι διαφημίσεις. Δηλαδή, αν έχετε μία στο, έναν ιστότοπο με ειδήσει. Όσο πιο πολλές ειδήσει έχει ο ιστότοπος αυτός, τόσο πιο πολλές διαφημίσεις θα λάβει. Και αυτό σημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι πιέζονται περισσότερο να παράγουν, να παράγουν ειδήσει. Και τώρα δεν έχουν να κάνουν μόνο ε, το άρθρο της εφημερίδας, αλλά έχουν να γράψουν και δύο-τρία άρθρα για την ε, Διαδικτυακή Ένωση, γιατί από αυτό εξαρτάται το εισόδημά τους. Αυτό που θέλω εγώ λοιπόν να ρωτήσω είναι, ο τρόπος που χρηματοδοτούνται οι εφημερίδες είναι και αυτό μήπως ένας παράγοντας Επίσης υπάρχει και η συνεχόμενη παροχή ε, και κάλυψη. Πολλά μέσα έχουν 24 ώρη κάλυψη ειδήσεων και αυτό δυσχεραίνει το έργο των ερευνητικών δημοσιογράφων. Άρα λοιπόν πρέπει να κοιτάξουμε και την ε, οργάνωση της δημοσιογραφίας καθ' αυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, Ίνες. Η κυρία Ινέσα Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λυπούμε, διότι δεν έφτασα εγκαίρος και δεν μπόρεσα να ακούσω τις εξηγήσεις. Ήμουνα στην Επιτροπή Μεταφορών και εκεί είχαμε ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα. Δεν συμφωνώ 100% με τον κύριο Ντόιτς Πιστεύω ότι και μόνο το γεγονός ότι έχει περιληφθεί τόσο πολλή δουλειά σε αυτή την έρευνα και τη μελέτη και μόνο το γεγονός ότι περιλαμβάνει συστάσεις σε τόσο δύσκολες στιγμές για, την, για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, το γραπτό τύπο και την οπτικοακουστική δημοσιογραφία και μόνο το ότι υπάρχουν όλα αυτά είναι μια ε, έντιμη προσπάθεια και θα πρέπει να εκφράσουμε την εκτίμησή μας για αυτή. Από εκεί και πέρα. Διατρέχουμε τον εξής πολύ σημαντικό κίνδυνο. Οι μεγάλοι όμιλοι τύπου πληροφόρησης δεν δίνουν προτεραιότητα στην ανεξάρτητη πληροφόρηση του κόσμου, δίνουν προτεραιότητα στην επιβίωση του στην οικονομική και στην εισαγωγή του στο χρηματιστήριο. Εξού και δημιουργούνται μονοπωλιακές καταστάσεις και γι' αυτό θέλουν να πουλήσουν ως θέμα τα πάντα ε, και να ε, πρημοδοτήσουν τα σκάνδαλα της ιδιωτικής ζωής του ενός και του αλουνού, ε, να πρημοδοτήσουν τα ποινικά θέματα και όλα αυτά τα σκανδαλοθυρικά θέματα που πουλάνε υποτίθεται περισσότερο. Αυτή τη στιγμή διανύουμε μια οικονομική, κοινωνική κρίση πολύ σημαντική και θα πρέπει να διαβάσει ο κόσμος περισσότερο για να μάθει την ισπανική πραγματικότητα, τη γερμανική πραγματικότητα. Ο ΜΕΝ πρέπει να διαβάζει την ε, επικαιρότητα και την πραγματικότητα του ΔΕ για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τους εαυτούς μας καλύτερα. Και ε, για να έχουμε σωστή ευρωπαϊκή διαχείριση της κρίσης και διακυβέρνηση και για να τα τα φέρουμε αυτά χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό τύπο, ευρωπαϊκά μέσα ε, μαζικής επικοινωνίας και όχι μέσα μαζικής επικοινωνίας που υπηρετούν εθνικά ε, συμφέροντα και που λειτουργούν οφειλημιστικά. Να μην σας θυμίσω το θέμα με τα ισπανικά αγκούρια ε, και με την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων στα σχολεία της Γερμανίας που υποτίθεται ότι αναφέρθηκε και λάθος ότι ήταν ισπανικής προέλευσης ενώ τελικά αποδείχθηκε ότι καμία σχέση. Χρειαζόμαστε λοιπόν περισσότερη διαχείριση, καλύτερη διακυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περισσότερη διαφάνεια ώστε να διευκολύνονται οι επαγγελματίες της ερευνητικής δημοσιογραφίας. Συν τις άλλες, χρειαζόμαστε ε, κώδικα δεοντολογίας. Το απαιτούμε και για την Όλαφ αυτό. Κώδικο δεοντολογίας για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα οποία πράγματι φυτοζωούν ενδεχομένως, έχουν υποστεί πάρα πολλές περικοπές, ε, κινδυνεύουν οι θέσεις τους και γι' αυτό ε, πολύ συχνά υποκύπτουν στον πειρασμό να κυτρινήσουν και να κινηθούν πιο πολύ προς την κίτρινη δημοσιογραφία. Ε, προτείνονται βέλτιστες πρακτικές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό στο κείμενο που έχουμε μπροστά μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο που σας ανέφερα μόλις τώρα και σύν της άλλης ε, με όλα αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με όλες τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας, του διαδικτύου, πολύ συχνά γίνονται πολύ πιο ευπαθείς συγκεκριμένοι θεσμοί, κάποιες ομάδες και πρέπει να δούμε ε, πώς θα καταφέρουμε να επιτύχουμε πάλι τον επαγγελματισμό, την ανεξαρτησία, τον τον πλουραλισμό και περισσότερη διαφάνεια για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην πληροφόρηση των ε, δημοσιογράφων που ασκούν ερευνητική δημοσιογραφία. Εάν ε, περιοριστεί το πεδίο δράσης της ερευνητικής δημοσιογραφίας, τότε η δημοκρατία θα δεχθεί ένα πολύ ισχυρό πλήγμα. Και όσο περισσότερο μπορούμε να δράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκεί, τόσο το καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφος Σάβαμεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ήμουν δημοσιογράφος επί 25 χρόνια και μέσα στα καθήκοντά μου ήταν και η ερευνητική δημοσιογραφία. Έχω λοιπόν και αυτό στο βιογραφικό μου. Θα ήθελα λοιπόν να θίξω κάποια σημεία. Νομίζω πως ο Δανός φίλος μας μας υπενθύμησε και καλά έκανε το τρίγωνο των Βερμούδων που υπάρχει. Όμως, εκείνος το παρουσίασε ως μία αρνητική ροή εξουσίας. Έναν φαύλο Εγώ προσωπικά το βλέπω, θα ήθελα να το δω διαφορετικά, θα ήθελα να το δω με θετικό πρόσημο. Οι δημοσιογράφοι, και το ξέρω αυτό εκ πείρας, ενδιαφέρονται για τέτοια για τέτοιες ειδήσει, για τέτοιες περιπτώσεις και πιστεύω πως εάν αυτές οι περιπτώσεις είχαν μεγαλύτερη κάλυψη αυτό θα ενδιαφέρε και το κοινό το να μάθουν τι γίνονται τα χρήματά τους. Και όσον αφορά το, τη μία αγωνία του τριγώνου, τους πολιτικούς, και οι πολιτικοί ενδιαφέρονται να μαθευτεί η αλήθεια. Το 99% από εμάς δεν έχει τίποτα να κρύψει. Υπάρχει λοιπόν, εγώ τουλάχιστον βλέπω ένα θετικό κύκλο και όχι ένα φαύλο κύκλο. Περίπου 3.000 άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονται στον κλάδο του τύπου. Πρέπει πραγματικά να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη και να αναλογιστούμε. Βοηθούμε τους δημοσιογράφους όπως θα έπρεπε. Και πολύ φοβάμαι πως όχι, σε καμία περίπτωση. Ας μην, λοιπόν, κρίνουμε μόνο αλλά ας δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να τους βοηθήσουμε. Πιστεύω πως η έκθεση περιλαμβάνει πάρα πολύ καλές συστάσεις και στα συμπεράσματα αναφέρονται πολύ σωστά πράγματα. Για παράδειγμα, τον, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την εστίαση σε αυτά που είναι πραγματικά σημαντικά. Δεν ξέρω αν με αντιλαμβάνεστε. Αλλά πιστεύω πως μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αλήθεια είναι ότι πολλές φορές, αρκετές φορές, οι δημοσιογράφοι ταμπελιάζουν. Αλλά ακόμα περισσότερες φορές είναι σαν τυφλοί που περπατούν στο δάσος. Τους πετάς ένα ξεροκόμματο και τους ενδιαφέρει και το κυνηγούν. Αλλά, όπως αναφέρεται και στην έκθεση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ένας μόνο ρεπόρτερ ή μία, ένα μόνο μικρό μέσο ενημέρωση να ασχοληθεί με άρθρα, με ειδήσει τόσο περίπλοκες, με θέματα τόσο μεγάλα. Χρειάζονται λοιπόν και βοήθεια από εμάς, τους ίδιους, και πιστεύω ότι αυτό θα μας πάει πολύ μπροστά. Σας ευχαριστώ και για μία ακόμα φορά συγχαρητήρια για την έκθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στάς. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο. Πολύ σωστά πράγματα αναφέρθηκαν. Η μελέτη αυτή τονίζει όντω την ανάγκη καλύτερη συνεργασίας μεταξύ δημοσιογράφων, διότι η διεθνή συνεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος αποκάλυψης γεγονότων. Ωστόσο, σε έναν ολόνα και περισσότερο ανταγωνιστικό κλάδο, τον κλάδο των μέσων ενημέρωσης. Πώς μπορούμε όταν όλοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους να συνεργαστούμε για να φέρουμε στο φως γεγονότα και να ανταλλάξουμε πληροφορίες. Πώς μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον ανταγωνισμό επικοδομητικό. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Έχουμε πρόβλημα χρόνου, δυστυχώς μέχρι τις 11 και 35. Γι' αυτό λοιπόν παρότι είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε θα ήθελα σας παρακαλώ να είστε σύντομοι και να αναφέρετε μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους για τις ερωτήσεις σας. Με χαρά μου διαπιστώνω ότι διαβάσατε και διεξοδικά μάλιστα την μελέτη. Είμαι ανοιχτή στην κριτική παρά το γεγονό ότι πολλοί, από εμάς δεν αντιδρούμε θετικά στην κριτική. Εγώ και ο κύριος Ντεμπρέιν θα απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας. Καταρχάς, ο πρώτος ε, ομιλητής είχε ορισμένα καλά σημεία, ο συνάδελφος από την Ουγγαρία. Με χαρά να σας απαντήσω κατηδίαν. Πράγματι, δώσαμε βάση σε ορισμένα διαδικτυακά μέσα όταν αναλύσαμε την κατάσταση στην Ουγγαρία. Ήθελα να ασχοληθώ και με άλλα, όμως έδωσα προσοχή στα διαδικτυακά μέσα, γιατί εκείνα είναι τα μέσα τα οποία ασχολούνται με ε, την απάτη στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπήρξαν πάνω από 100 άρθρα τα τελευταία πέντε χρόνια. Αυτό όμως ε, που εμείς ε, θέλαμε να τονίσουμε είναι την ερευνητική δημοσιογραφία, διότι πραγματικά θέλαμε να αναλύσουμε εις βάθος το τι κάνουν οι δημοσιογράφοι από μόνοι τους, τι ξεθάβουν από μόνοι τους και όχι τι τους δίνεται. Και θέλαμε λοιπόν γι' αυτό να δούμε ποια μέσα, ηλεκτρονικά ή μη, ασχολούνται με ακριβώς αυτό το πράγμα, το να φέρνουν στο φως καινούργια στοιχεία. Και όσον αφορά την κριτική που ασκήθηκε για τον νόμο για τα μέσα ενημέρωση στην Ουγγαρία, ναι, ήταν αναμενόμενο. Και αυτό που μας είπαν ε, από την ουγγρική πλευρά είναι ότι δεν παρεμποδίζει τη δουλειά των δημοσιογράφων. Οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με την ερευνητική δημοσιογραφία πάντως είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν το έργο τους και δεν θεωρούν τον νέο, νόμο, τον νέο Ουγγρικό νόμο για τα μέσα ενημέρωσης εμπόδιο, παρότι μπορεί να μην βοηθά γενικά τον δημοσιογραφικό κλάδο. Ένα αίτημα από τον πανεπιστημιακό χώρο ήταν να γίνει μια συνολική συνοπτική θεώρηση των, ε, της νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης στην Ευρώπη των 27 και όχι να ασκήσουμε κριτική ή να επικροτήσουμε τη συμπεριφορά ορισμένων χωρών, αλλά να κάνουμε μια γενικότερη συνοπτική θεώρηση της συμπεριφοράς της ε, νομοθεσίας για τα μέσα ενημέρωσης. Και πραγματικά πιστεύω πως ε, η έρευνα για τις βέλτιστες πρακτικές στην ε, δημοσιογραφική νομοθεσία θα ήταν πάρα πολύ σημαντική και θα μας βοηθούσε, θα ήταν μια συγκριτική αξιολόγηση. Η και ο συνάδελφο που εκπρόσωπευε την ε, αντίστοιχη Ουγγρική Αρχή μα είπε ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Τώρα, οι δύο ευρωβουλευτέ από την Πολωνία. Να, καταρχάς να σας ευχαριστήσω. Θίξατε ένα πολύ σημαντικό θέμα, τον πατριωτισμό ή την κριτική δημοσιογραφία. Είναι πολύ δύσκολο ζήτημα και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε περιπτώσεις όπου δημοσιογράφοι ασκούν κριτική στον στο κράτος, διότι πολλοί φοβούνται ότι εάν ασκήσουμε κριτική, του χρόνου δεν θα έχουμε κονδύλια. Σας ευχαριστώ λοιπόν που θίξατε το ζήτημα αυτό. Είναι κάτι που πρέπει ως δημοσιογράφοι να έχουμε υπόψη. δεν σημαίνει. Ε, όσον αφορά τον συνάδελφο από το Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, δεν σημαίνει ότι κάθε Βρετανό δημοσιογράφο είναι ευρωσκεπτικιστή ή κάθε ε, υπάλληλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φιλοευρωπαίο. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η μεροληψία. Γι' αυτό χρειάζεται και εξάλλου διαφάνεια. Πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη. Διαφορετικά κινδυνεύουμε να γίνουμε ως νοσογράφοι πιόνι. Και αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να μας συμβεί. Να γίνουμε δηλαδή πιόνια οποιασδήποτε από τις δύο πλευρές. Επίσης εδώ αναφέρθηκε κάτι που ανέφεραν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Τα, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ανεξάρτητα μέσα, ανεξαρτησία του τύπου. Και από τις έρευνές μας έρευνές μας καταλήξαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά μικρά μέσα ενημέρωσης που ασχολούνται με την ερευνητική δημοσιογραφία, τα οποία δεν λαμβάνουν καμία χρηματοδότηση και αυτά χρειάζεται να βοηθηθούν. Τώρα, υπήρξαν αρκετά ερωτήματα για την προστασία των δημοσιογράφων. Εμείς αυτό που βρήκαμε από τις μελέτες μας είναι ότι πρέπει να προστατεύσουμε την δημοσιογραφική διαδικασία και όχι τους ίδιους τους δημοσιογράφους. Εάν μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία και την ασφάλεια της δημοσιογραφικής διαδικασίας, τότε ως επακόλουθο θα υπάρξουν και δημοσιογράφοι που θα κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Ξέρω ότι η έννοια της ε, προστασίας της δημοσιογραφικής διαδικασίας ακούγεται κάποιο, κάπως αφηρημένη, όμως και αυτό θα οδηγήσει στο ποιος είναι δημοσιογράφος και ποιος όχι. Ή το ποιος μπορεί να έχει προστασία ή όχι. Πρέπει πραγματικά να δούμε την διαδικασία και αυτή να προστατεύσουμε και εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό. Η κυρία Σαραντίνη ανέφερε την πρόσβαση στα έγγραφα και το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε το ισχύον καθεστώς. Αυτό που θα προτείναμε εμείς είναι να κοιτάξετε τις βέλτιστες πρακτικές σε ορισμένα κρατημέλη, υποδείγματα. Κάποια κρατημέλη όπως το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν καθυστερήσει στην εφαρμογή της ελευθερίας του τύπου. Όμως, τώρα έχουν δείξει μεγάλο ζήλο και βοηθούν τους δημοσιογράφους να έχουν ε, εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα. Γι' αυτό πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει το να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές ανά κράτος μέλος. Γνωρίζω πως η Δανική Προεδρία για τους, τελευταίους 6, για τους πρώτους 6 μήνες του 2012 εργάστηκε πάνω σε αυτό. Και νομίζω πως αυτό είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε και κατηδίαν. Θα θέλαμε να το σκεφτούμε λίγο και να σας δώσουμε ορισμένε κατευθυντήριες γραμμές. Ευχαριστώ, ο κύριος Δεμπρέν με τώρα. Ο κύριος Δεμπρέν, λοιπόν, θα ήθελα να σας πω το εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον προσπαθεί να μιλήσει για τη διαφάνεια της ε, δημόσιας διοίκησης και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι απαραίτητο. Η κυρία Σαρτζεντίνη στην ε, παρέμβασή της μίλησε για τον πλουραλισμό των μίντια, πώς μπορούμε να τον ενθαρρύνουμε και να τον αναπτύξουμε. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη βάση του θέματος πώς θα ενισχύσουμε το πλουραλισμό αλλά και την ερευνητική δημοσιογραφία γενικότερα. Νομίζω ότι οι ίδιοι δημοσιογράφοι πρέπει να καταρτήσουν νέο επιχειρησιακό σχέδιο. Δηλαδή, με τις διαδικτυακές δημοσιεύσεις τους να δημιουργήσουν τα δικά τους δίκτυα. Και γι' αυτό είναι και πολύ σημαντικό ο ΦΠΑ πάνω στις ε, στις ε, διαδικτυακές δημοσιεύσεις, αν θα είναι χαμηλός ή υψηλός και πώς θα ενισχύσουμε αυτή την ερευνητική δημοσιογραφία και πώς θα επιτρέψουμε στο δημοσιογράφο να προστατεύσει τις πηγές του. Τι πρέπει να κάνει ένας δημοσιογράφος για να ερευνά. Ε, πρέπει να έχει χρόνο, πρέπει να είναι παρόν. Άρα πρέπει να χαίρει υποτροφιών από ιδρύματα όπως τα δικά μας έχουμε το journalistfund.eu. Εκεί οι δημοσιογράφοι μπορούν να έχουν υποτροφίες για διασυνεωριακή συνεργασία. Δυστυχώς, σήμερα στην Ευρώπη δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα ε, για όλα αυτά. Πρέπει να πείσουμε λοιπόν τα ευρωπαϊκά ιδρύματα να βοηθήσουν. Και είναι πολύ λεπτό το ζήτημα, ε, γιατί πολύ σπάνια χρηματοδοτούνται οι δημοσιογράφοι. Πώς θα ενθαρρύνουμε τους δημοσιογράφους χωρίς να ενθαρρύνουμε τα μίντια. Τα μίντια. Ευχαριστώ. Πράγματι, τα μίντια είναι επιχειρήσεις. Ε, σχολιάζει η επόμενη ομιλήτρια. Και αυτό είναι πρόβλημα. Εάν όμως ε, κοιτάξουμε το πώς θα σώσουμε τη δημοσιογραφία και όχι την εφημερίδα, τότε θα κάνουμε καλή δουλειά. Πολύ συχνά ορισμένες εφημερίδες δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Το διαδίκτυο είναι πολύ πιο γρήγορο. Ωστόσο, άλλες φορές ε, έντυπα που εστιάζουν την προσοχή τους στην ερευνητική δημοσιογραφία αποκτούν όλο και πιο ισχυρές βάσεις. Σιγά σιγά διεισδύουν περισσότερο γιατί τελικά ο κόσμος θέλει να διαβάσει ε, καλή δημοσιογραφία, ένα καλό δημοσιογραφικό άρθρο. Μου τέθηκε και ερώτημα για το ρόλο των δημοσιογράφων και τη στήριξή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πράγματι, το λάβαμε υπόψη μας. Και γι' αυτό έχουμε και το σχέδιο του Γραφείου για την Ερευνητική Δημοσιογραφία. Πολύ συχνά χρειάζεσαι έναν εξωτερικό συνεργάτη για να κάνει τέτοιου είδου έρευνε, γιατί ο τύπο είναι τόσο διαιρεμένο και τόσο πολιτικοποιημένο ή κομματικοποιημένο, που μόνο τη μία πλευρά τη ιστορία θα μάθει εάν αναθέσει αυτήν την ερευνητική δουλειά σε συγκεκριμένο δημοσιογραφικό όμιλο ή ενημερωτικό όμιλο. Γι' αυτό και είπα εγώ εξ αρχή όσο πιο πολύ, τόσο πιο καλά. Όσο περισσότερο πλουραλισμό, τόσο περισσότερη ανεξαρτησία στην ερευνητική δημοσιογραφία πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν να τους προσεγγίσουμε αυτούς τους ανεξάρτητους ερευνητές δημοσιογράφους που έχουν πολλά να προσφέρουν. Ο κύριος από τη Γερμανία με ρώτησε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την παροχή των στοιχείων προς τα κράτη-μέλη, πώς αξιολογεί τη στάση της. Καλά τα πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη είναι το πρόβλημα. Δηλαδή τα κράτη-μέλη όταν δίνουν στοιχεία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, εκεί υπάρχει περισσότερο πρόβλημα στην πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Η ομοιόμορφη συγκέντρωση, η συλλογή δεδομένων αριθμητικών στοιχείων είναι πραγματικά το α και το ω. Και πώς θα αναδιαρθρώσουμε το 2% των κονδαλίων, των 18 εκατομμυρίων δολαρίων που αναφέρθηκαν στην έκθεση ΣΥΜΑ, το 2% που πηγαίνει για την ερευνητική δημοσιογραφία. Κοιτάξτε, Πάρα πολλά χρήματα δαπανώνται σε αυτό που είπε και η κυρία Αγιάλα. Πανευρωπαϊκός πανευρωπαϊκή δημοσιογραφία. Δεν έχουμε μια πανευρωπαϊκή ε, εφημερίδα. Τη χρειαζόμαστε όμως. Ενδεχομένως όχι. Θα μπορούσε κανείς να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό κέντρο ερευνητικής δημοσιογραφίας. Αυτό το λέμε στην έκθεση κάνει την έρευνα μία φορά και τη δημοσιεύει 27 φορές, γιατί κάθε χρόνο αναδημοσιεύει τα στοιχεία που την αφορούν εκείνη προσωπικά. Κάνουμε την έρευνα άπαξ και μετά κάνουμε τη διάδοση των αποτελεσμάτων παντού. Έχουμε και την ευρωπαϊκή δημοσιογραφία, όχι τα ευρωπαϊκά μίντια, την ευρωπαϊκή δημοσιογραφία ως έννοια. Τα κέντρα εκεί μπορούν να διαδραματίσουν ένα πολύ σημαντικό ε, ρόλο. Και ένα τελευταίο νομίζω ε, που θέλετε να σχολιάσω. Ναι, ο κύριος Στάς μας είπε ότι σε ένα πιο, όλο και πιο ανταγωνιστικό μηντιακό τοπίο πώς πείθετε τους δημοσιογράφους να συνεργαστούν και να μην ανταγωνιστούν ο μεν τον δε μόνο όταν δουλεύουμε διασυνοριακά. Δηλαδή αν δουλεύει κανείς στη Μαδρίτη σίγουρα ε, ε, το συναδέλφό του από τη Λετωνία δεν τον βλέπει ανταγωνιστικά. Είναι ο, ο κάθε ένας για τον άλλον αποτελεί στοιχείο ενεργητικού και όχι παθητικού. Εξού και εκεί μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δημοσιογραφία. Ποτέ κανεί δεν βρίσκει ανταγωνιστή και δεν έχει να αντιμετωπίσει αδυσόπιτο ανταγωνισμό όταν εργάζεται διασυνοριακά. Σίγουρα η εσωτερική συνεργασία εντό τη ίδια χώρα είναι πιο δύσκολη. Αλλά θα μπορούσε για παράδειγμα οι δημοσιογράφοι τηλεοπτικού σταθμού να συνεργάζονται με δημοσιογράφου εφημερίδα ή με δημοσιογράφου κάποια διαδικτυακή τοποθεσία. Είναι κάτι που έχει συμβεί, που συμβαίνει, που το δείχνουμε στο γραφείο ε, της ε, δημοσιογραφίας της ερευνητικής. Το Al Jazeera συνεργάστηκε το κανάλι με το ε, ραδιοφωνικό κανάλι του BBC, το BBC Radio και πήγαν πολύ καλά τα πράγματα. Αυτά προς το παρόν ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρατήρηση. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι λιγότερο περίπλοκη. Δεν νομίζω ότι πρέπει τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να είναι λιγότερο περίπλοκα. Αυτό που πρέπει είναι να διευκολύνουν τους δημοσιογράφους να εξηγούν την περιπλοκότητα, να κάνουν τα πράγματα πιο απλά, να εξηγούν ποιες είναι οι λανθάνωσες, οι αποχρώσεις έννοιες αυτές, αυτής της πολυπλοκότητας για να τις καταλαβαίνουν καλύτερα οι δημοσιογράφοι και να μπορούν να τις αναμεταδώσουν. Το σημαντικό είναι ότι οι δημοσιογράφοι θα πρέπει να κατανοήσουν την περιπλοκότητα των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να μπορέσουν να την εξηγήσουν καλύτερα και στην κοινή γνώμη. Νομίζω λοιπόν ότι με αυτά έχουμε ε, ολοκληρώσει ε, τις απαντήσεις. Ε, κύριε Σμιτ, κάνατε το παν για να απαντήσετε στις ερωτήσεις εντός του προκαθορισμένου χρόνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελειώνω, λοιπόν ο συνάδελφος ε, Μπάστας ε, ως εισηγητής. Κοιτάξτε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Ε, καταρχήν θέλω να πω ότι κατά την άποψή μου είναι σημαντικό να διαδώσουμε περαιτέρω αυτή την έκθεση. Εχθές πήραν τη μελέτη και Επίτροπος κ. Σεμέτα και ο Επίτροπος Κρούς και νομίζω ότι ε, καλό είναι αυτό γιατί η έκθεση αυτή αφορά και ορισμένα μέσα της ενημέρωσης. Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα από την έκθεση αυτή. Εμείς ε, ως ε, θεσμοί οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι οποτεδήποτε έρχονται οι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί. Η διαφάνεια των δραστηριοτήτων και κατά τη λήψη αποφάσεων, η καλύτερη διαχείριση των στοιχείων το απόρριτο των στοιχείων, η καλύτερη προστασία των πηγών, των δημοσιογράφων και η ε, προστασία της διασυνοριακής συνεργασίας ε, δημοσιογράφων. Αυτά τα στοιχεία στη σημερινή εποχή, την εποχή του ανταγωνισμού, είναι πάρα πολύ σημαντικά δημοσιογράφοι βεβαίως ε, είναι στη διάθεσή σας ε, εφόσον ε, θέλετε να τους υποβάλλετε και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμφωνώ και παυξάνω, λέει ο Πρόεδρος. Τέτοιου είδου συζήτηση δεν είχαμε εδώ και πολύ καιρό. Ευχαριστούμε τον Μάρκο Βίτ και την Ίντεστε Μπρουίν για την εκπόνηση αυτής της μελέτης. Κλείνει αυτό το σημείο της σημερινής διάταξης και πάμε στο επόμενο όπου η συγγήτρια είναι η Εύα Ορτής Βιλέλα. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Βούγκεπάουα να κάνει την εισαγωγή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα μπορώ να σας παρουσιάσω την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη μεταρρύθμιση της κοινή οργάνωσης αγοράς στον αμπελονικό τομέα. Να σας παρουσιάσω την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα και επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να κερδίσουμε λίγο χρόνο ε, Ε, πρέπει να ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στον τομέα αυτό και παράλληλα η παραγωγή ίνου ε, είναι το 5%. Ε, το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι υφίσταται συνεχής ανισορροπία ανάμεσα στην παραγωγή και τη ζήτηση. Είχαμε ένα μεγάλο πλεόνασμα. Το 2011 είχαμε 50 εκατομμύρια ε, πλεόνασμα, λίτρα είναι αυτά πάντα. Και ε, αυτά με βάση τον ε, κανονισμό του 2008, όπου προβλέπεται η προαγωγή των μέτρων εκρίζωσης, αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας. Το θέμα είναι το εξής, το, η ζήτηση εδώ και 20 χρόνια πέφτει η κατανάλωση κρασιού μειώνεται διότι έχουν αλλάξει οι συνήθειες ε, κυρίως ε, ε, στις νότιες χώρες. Πολλοί αφήνουν το κρασί και πάνε στο νερό, στην πύρα, στα μη εινοπνευματώδη Αυτό καλό είναι για την υγεία, Άρα δηλαδή υπάρχει αυτό το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στο μέλλον. Υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα. Σε κάποια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται η κατανάλωση και αυτή η κατανάλωση ε, καλύπτεται όμως όλο και περισσότερο από εισαγωγές από τρίτες χώρες. Έχουμε πολύ καλούς ε, παραγωγούς ε, από τρίτες χώρες που παράγουν κρασί μεσαίας ποιότητας και χαμηλής ποιότητας και βρίσκουν όμως τα προϊόντα του ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα δηλαδή ο στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ανισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση. Το 2005 είχαμε ε, πλεόνασμα 14,5 εκατόλιτρα και στην απόσταξη 18,5 εκατομμύρια εκατόλιτρα. Το 2008 ε, είχαμε 4 δις ευρώ έσοδα. Τα σημαντικότερα μέτρα τα είπα, το πριμ, η πριμοδότηση της εκρίζωσης που υπήρχε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά με τον καινούριο κανονισμό κρασιού το 2008 έλαβε μια νέα μορφή. Όσοι λοιπόν είχαν τέτοιου είδους επιχειρήσεις και όσοι έχουν μπορούν να ζητήσουν ε, επιδότηση και αυτή η αλλαγή αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Η πλημοδότηση το πρώτο χρόνο αυξήθηκε κατά 20%, το δεύτερο 10% και τον τρίτο χρόνο παραμένει στο ίδιο επίπεδο όπως και κατά το παρελθόν. Μετά από τρία χρόνια, το 8 έως 10, το ύψος των διατηθέμενων κονδυλίων ε, που μπορούσαν να προσφερθούν για τέτοιου αιτήσει ε, ξεπεράστηκε. Τώρα, η μείωση η οποία αναμένεται δεν έφτασε, δεν φτάσαμε σε αυτή τη ε, μείωση. Ε, υπήρξε ένα μεγάλο μεγαλύτερο ποσό που ε, ζητήθηκε, αλλά φτάσαμε σε 160.000 περίπου ε, εκτάρια εκρίζωσης. που αντιστοιχούσε σε περίπου 6% της ε, παραγωγής. Πάω τώρα στο δεύτερο θέμα, στα μέτρα, στην αναδιάρθρωση των ε, των αμπελώνων. Το μέτρο αυτό υπήρχε ήδη πολύ πριν εισαχθεί ο νέος κανονισμός αγοράς κρασιού το 2008. Τα μέσα ήταν 4,2 ευρώ ε, το 2001 στο 2010, δηλαδή 420 ε, εκατομμύρια το χρόνο. Το ποσοστό ε, στο σύνολο των κονδυλίων της μεταρρύθμισης 32%. Στόχος αυτού του μέτρου ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από την αναδιάταξη, αν διάταξη των αμπελώνων και νέες ε, τακτικές και ε, τεχνολογίες διαχείρισης. Επίσης ε, να υπάρξει αποζημίωση του εισοδήματος κατά τη διάρκεια της προσαρμογής και επιδοτήσεις για το κόστος αναδιάρθρωσης. Εδώ λοιπόν θέλω να σας επισημάνω κάτι πολύ σημαντικό, δηλαδή ε, το κόστος αναδιάρθρωσης και αναπροσαρμογής ε, στα κράτη-μέλη έφτασε ε, μέχρι 200% ανά εκτάριο. Καταλαβαίνετε αυτό ήταν παράλογο διότι ειδικά σε κράτη όπου το κόστος εργασίας είναι πολύ χαμηλό εκεί η υπήρχε μεγαλύτερο κόστος αναδιάρθρωσης από τις σε χώρες που είχαν ε, υψηλό κόστος εργασίας. Παράδειγμα συγκεκριμένο, Ρουμανία. 200% υψηλότερο κόστος ε, αναπροσαρμογής από τη Γερμανία, παρότι ε, το κόστος εργασίας ε, στην ε, Ρουμανία δεν μπορεί να είναι τόσο υψηλότερο από τη Γερμανία. Οι επιπτώσει από αυτό το κόστος αναπροσαρμογής και αναδιάρθρωσης, αυτές μπορώ να, σα να σας δείξω με δύο παραδείγματα. Στην Καστήλια Λαμάντσα, το 16% τα τελευταία 10 χρόνια αναδιαρθρώθηκε στο Λόγκτο Κροσινιό, το 21%. Το πρόβλημα λοιπόν ε, προκύπτει ω εξή. Η αύξηση της απόδοσης είναι εκείνη η οποία καταστρέφει ε, εν μέρη και συχνά πλήρως ε, το όφελος της εκρίζωσης. Και πάλι δύο παραδείγματα. Στην Ισπανία υπήρχε αύξηση απόδοσης 50 εκατομμύρια εκατόλιτρα και αυτή η αύξηση της απόδοσης ήταν κατά 13% μεγαλύτερη από την μείωση λόγω των εκριζώσεων. Τώρα, ε, στην Καστήλια Λαμάντσα οι εκτάσεις που εκρυζώθηκαν ήταν κατά 60% 40% υψηλότερες από εκτάσεις που δεν αναδιαρθρώθηκαν. Η ανάλυση της συγκομιδής ε, δείχνει ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχει ε, σημαντική αύξηση της ε, παραγωγής. Και εδώ θέλω να σας παραπέμψω στο γράφημα υπαριθμό 1 στη σελίδα 9. Εκεί βλέπουμε ότι περίπου 30 εκατομμύρια εκατόλιτρα θα μπορούσε να είναι η επιπρόσθετη παραγωγή εάν ορισμένα κράτη-μέλη που δεν εμφανίζουν παραγωγικότητα ε, όπως ε, τα κράτη που έχουν υψηλή παραγωγικότητα, αν αυτά δηλαδή που δεν είναι παραγωγικά επιτύχαναν την ίδια παραγωγικότητα με τα άλλα. Και η αύξηση τους ε, παραγωγής θα ανήρχεται σε 20% στο μέλλον εάν οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκταμιευτούν. Άρα δηλαδή στα μέτρα που θα ληφθούν υπόψη αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου. Κατά τα άλλα, ένα πράγμα θέλω να πω ως αποτέλεσμα, εάν τελικά δεν υπάρχουν επιπρόσθετες δυνατότητες πώληση ε, για την αύξηση της παραγωγής που θα προκύψει μέσα από την αναδιάρθρωση, τότε το πρόβλημα των πλεονασμάτων θα είναι ακόμα χειρότερο. Και κάτι άλλο, τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξε μείωση, ε, όπως τα τελευταία 20 χρόνια, της κατανάλωσης. Οι εξαγωγές κρασιού ευτυχώς αυξήθηκαν κατά τη και γι' αυτό το λόγο ε, μειώθηκαν κατά τη πάλι οι αμπελώνες. Όμως από αυτές τις παρατηρήσεις δεν μπορούμε να εξάγουμε μακροπρόθεσμα συμπεράσματα και τούτο διότι προφανώς η παραγωγή κρασιού εξαρτάται από τον καιρό. Το 2011 είχαμε κακή συγκομιδή. Οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτώνται και από τις εξαγωγές κρασιού σε τρίτες χώρες. Στο ίδιο χρονικό διάστημα σε κάποια κράτη υπήρχε κακή συγκομιδή. Και ένα πράγμα δεν πρέπει να ξεχνάμε. Στην παγκόσμια αγορά κρασιού ρόλο, ρόλο οι ισοτιμίες. Αυτά τα τρία χρόνια λοιπόν που εξετάζουμε για κάποιες τρίτες χώρες υπήρξαν αρνητικές εξελίξεις στη συναλλαγματική αγορά που για μας σημαίνει ανατίμηση. Ε, τώρα, όσον αφορά τις συστάσεις, οι εκριζώσεις, η Κομισιόν με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν και ε, συμπεριλαμβανομένης ε, και της απελευθέρωσης των δικαιωμάτων φύτευσης θα πρέπει να αποφασίσει κατά πόσον και εάν πρέπει να ληφθούν ποια μέτρα για την άρση ενδεχόμενων ανισορροπιών. Τώρα θα αναφερθώ σε ένα πολιτικά πολύ ευαίσθητο θέμα, στα δικαιώματα φύτευσης. Η κατάργηση προβλέπεται για το 2010, μετά είχε προβλεφτεί, μετά αναβλήθηκε για το 2015 και ορισμένα κράτη μπορούν να ζητήσουν την μετάθεση μέχρι το 2018. Όμως εμείς συστήνουμε, επειδή δεν υπάρχει τελική αξιολόγηση των πλεονασμάτων από την κατάργηση αυτού του μέτρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε αξιολόγηση ανάλυση. Ο Επίτροπος κύριος Τσόλος ε, ήδη αντέδρασε, χαίρομαι πάρα πολύ τον Απρίλιο του 2002 ε, είχε συστήσει μια ομάδα εργασία και από τις εκθέσεις που έχω στη διάθεσή μου συνάγω ότι υπήρξαν ουσιαστικές συζητήσεις, άρα δηλαδή μπορεί να υπάρξει κάποια προσέγγιση εάν συνεχιστούν οι εργασίες όπως ακριβώς συνέβη κατά τις τρει πρώτες συνεδριάσεις. Και χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η ομάδα εργασία που συστήθηκε μάλλον το 2012 όπως ακριβώς το πρότεινε ο Επίτροπος. Και κάτι άλλο, αν κρυθούν απαραίτητα. Περαιτέρω μέτρα εκρίζωσης, τα κριτήρια πρόθεσης ε, θα πρέπει να εξετάσουν όχι μόνο τις επιχειρήσεις, αλλά και τις ε, εκτάσεις ε, υποεκρίζωση. Εμείς λοιπόν βρήκαμε τέτοια παραδείγματα, παραδείγματος χάρη μία ε, παραγωγή για κόκκινο κρασί, τεμπρανίλο, 420.000 ε, ευρώ επιδότηση και αυτός ο αμπελώνας όμως εκριζώθηκε. Άλλα παραδείγματα για την αναδιάρθρωση. Ο σαφής ορισμός ε, των επιδοτούμενων εκτάσεων, αυτό δεν ε, είναι καταληκτικό γιατί υπάρχουν κάποιες εκτάσεις που ορίστηκαν υπό αλλά δεν θα πρέπει να εκριζωθούν. Παραδείγματο χάνει στη Τσεχία η προστασία ε, των ζώων ε, προήχθη, επιδοτήθηκε με 300 ώρες. Αυτό επίμαχο, φιλεγόμενο το αποτέλεσμα. Κάτι άλλο, αν τελικά ε, η εκρίζωση βασιστεί σε καταπεκοπή ποσό ανά εκτάριο, τότε τα κράτη-μέλη θα πρέπει ε, να προσέξουν το κόστος το κόστος ε, για συγκρίσιμες ενέργειες ε, το έχω αναφέρει. Είδαμε ότι υπάρχουν αποκλήσεις μέχρι και 200% ακόμα και με την ίδια πυκνότητα ε, του αμπελώνα. Ενώ σας είπα ότι το κόστος εργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πολύ χαμηλότερο από άλλες. Άρα δηλαδή και εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να είναι πολύ προσεκτική όσον αφορά αυτή την κατάσταση. Τώρα, για το μέλλον, η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του κανονισμού αγοράς του 2008 ε, διέθεσε δισεκατομμύρια. Αποτέλεσμα ανισορροπία ανάμεσα στη ζήτηση και την προσφορά και παρέμεινε ίδια η κατάσταση. Άρα δηλαδή ο στόχος δεν, επι, δεν επιτεύχθηκε. Υπάρχει ζήτηση που οδηγεί σε όλο και επιδεινούμενη κατάσταση για την, στην προσφορά και τη ζήτηση, πρόβλημα με την παραγωγικότητα, Ρουμανία, Ισπανία, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στο γράφημα υπαριθμών 1 στη σελίδα 20 λοιπόν, το είπα ήδη, οφείλει να αξιολογήσει κατά πόσο είναι δυνατόν να υπάρξει αύξηση ε, της παραγωγής εάν απελευθερωθούν τα δικαιώματα φύτευσης. Αυτή όμως είναι μια πολιτική απόφαση. Αυτή τη στιγμή ε, πρόκειται να ε, εκπνεύσει η επιδότηση της απόσταξης που και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής. Οι τρίτες χώρες γίνονται ανταγωνιστικότερες όχι μόνο στην τιμή αλλά και στην ποιότητα. Βεβαίως και πρέπει να συνεχίζουμε να επιλέγουμε την ποιότητα όμως πρέπει επίσης να έχουμε κατά νου ότι το κρασί μεσαία τιμής και τα φτηνά κρασιά αυτά δεν πρέπει να πέσουν ε, απολύτω ε, στα χέρια των τρίτων χωρών, κυρίω στα σούπερ μάρκετ, κάτι που υπάρχει όμω αυτή τη στιγμή και είναι μια τάση που όλο επιτείνεται, άρα δηλαδή εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει κάποια μέτρα. Άλλο πρόβλημα, η προαγωγή του διαφημίσεων κρασιού δεν επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή ε, μπορούν σε τρίτε χώρε να κάνουν διαφήμιση, αλλά όχι σε βασικά βασικές χώρε εισαγωγή, όπω τη Μεγάλη Βρετανία, τη Σουηδία και σε άλλε σκανδιναβικέ χώρε. Κατόπιν τούτου, για να επιτευχθεί ο βασικότερος στόχο τη μεταρρύθμισης, που είναι να υπάρχει καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση, εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα σωστό μείγμα μέτρων. Η αντίφαση ανάμεσα στην εκρίζωση και από την άλλη η αύξηση της απόδοσης λόγω της αναδιάρθρωσης είναι λάθος. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσοχή σας και εμείς για το ότι συνοψίσατε τα αποτελέσματα από την έκθεση του Ελληνικτικού Συνεδρίου και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο για αυτή την έκθεση στην ε, συγγήτρια ε, Εύα Όρτη Σιμπιλέλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για την ε, έκθεση για τη μεταρρύθμιση στον αμπελοενικό τομέα, έναν κλάδο πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια έκθεση και μια έρευνα η οποία λαμβάνει υπόψη τις πολιτισμικές διαστάσεις στην κάθε χώρα. Η τελευταία μεταρρύθμιση έλαβε χώρα το 2007 και θα έχουμε καινούργια μεταρρύθμιση και που μάλλον μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει και πάλι το συμπεφωνηθέν και θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας διευκρινίσει τα πράγματα εδώ. Στην έκθεση λοιπόν λαμβάνεται υπόψη η επίκριση του ελεκτικού συνεδρίου, ότι δηλαδή οι περικοπές παραγωγής που περιμέναμε ουσιαστικά αντισταθμίζονται με τα άλλα μέτρα που είναι η αδιάρθρωση και η μετατροπή. Και άρα το Συμβούλιο Υπουργών ε, δέχθηκε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέτρο αυτό, το οποίο τελικά συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγής και έτσι δεν έχουμε το όφελος της μείωσης της παραγωγής που θέλαμε τελικά. Η ερμηνεία είναι εξαιρετικά ευρεία και δεν υπάρχει αρκετή αντιστάθμευση με συγκεκριμένες δράσεις. Αν θα έπρεπε να υιοθετήσουμε ε, την εκρίζωση, πρέπει να αποφύγουμε την εκρίζωση των εξυγχρονισμένων αμπελώνων, ε, για να μην υπάρχουν και προβλήματα ερμηνείας το κράτος μέλος θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε οι ενισχύσεις να μην ξεπερνούν τελικά τα πραγματικά έξοδα και δαπάνες που έχει κάνει ο παραγωγός. Έχουμε τη μελέτη του αντικτύπου για την απόφαση κατάργηση των δικαιωμάτων φύτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προτείνεται να γίνεται εκ των προτέρων αξιολόγηση. Θα ήθελα λοιπόν να υπενθυμίσω τη θέση των 16 κρατών μελών υπέρ της ε, αναθεώρησης της απόφασης του 2007 για την κατάργηση των δικαιωμάτων φύτευσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φρονεί το ίδιο και το έχει πει επανειλημμένος ότι στη συζήτηση για τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής η έκθεση του βουλευτή Άλμπερτες την περασμένη χρονιά ως προς τη μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής ζήτησε τη διατήρηση των δικαιωμάτων φύτευσης και μάλιστα το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Μίτσελ Λάντιν για την κοινή οργάνωση ε, αγοράς για τα γεωργικά προϊόντα ε, ζητά την παράταση αυτών των δικαιωμάτων μέχρι το 2030. Και αυτό την χάνει ευρεία υποστήριξη ε, μεταξύ των συναδέλφων μα στην Επιτροπή Γεωργία. Είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για αυτό το θέμα αυτό σήμερα, διότι έχει να κάνει με την ισορροπία μεταξύ ε, ζήτηση και προσφορά, που είναι το ζητούμενο σε αυτό το κλάδο. Επομένω, δεν θα πρέπει να πάρουμε απόφαση λάθο εστιασμένη, λάθο ζυγιασμένη και θα πρέπει να ε, εξαλείψουμε τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα, ακριβώς διότι έχουν, έχουμε θετική εξέλιξη στις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Με την τελευταία μεταρρύθμιση έχουν επιτευχθεί σημαντικά, έχουν γίνει σημαντικά βήματα και δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Η εκρίζωση και οι ενισχύσεις έχουν οδηγήσει ε, σε ε, αποτελέσματα. Καμία μεταρρύθμιση δεν είναι τέλεια, αλλά από το 2010 και μετά έχουν, ε, σημειώνουν άνοδο οι εξαγωγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο αντισταθμίζει την πτώση της κατανάλωσης στις χώρες παραγωγούς. Στην έκθεσή μου λοιπόν τονίζω πόσο ανταγκαίο είναι σε θέματα κρασιού η ευρωπαϊκή πολιτική στο μέλλον να μην περιλαμβάνει τίποτα το αντιφατικό. Εάν για να πετύχουμε τους ε, στόχους μας θέλουμε να βελτιώσουμε την αναδιάρθρωση των αμπελώνων, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να μελετήσει σε βάθος πώς θα βελτιώσουμε τις δράσεις μας για να είναι πιο ανταγωνιστικός ο τομέας. Και βεβαίως πιστεύω ότι η πολιτική αναδιάρθρωση των αμπελώνων δεν θα πρέπει να συνδυάζεται με μέτρα που οδηγούν οδηγούν τελικά σε ανισορροπίες στην προσφορά και τη ζήτηση. Και αυτό κατά τη γνώμη μου θα συμβεί εάν καταργηθούν τα δικαιώματα φύτευσης και απελευθερωθούν τελικά. Και θα πρέπει να ενισχύσουμε την προώθηση του ευρωπαϊκού κρασιού στην εσωτερική αγορά, να έχουμε εκστρατείες ενημέρωσης πληροφόρησης για την αξία των ευρωπαϊκών κρασιών, ούτω ώστε να ενισχυθεί η εσωτερική κατανάλωση. Πάντοτε βεβαίως με την ε, έκκληση για υπεύθυνη και ε, περιορισμένη κατανάλωση για λόγους υγείας, μεταξύ άλλων. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει ενισχύσιμο μέτρο σε εσωτερικό επίπεδο, ενώ από την άλλη, ε, διακόπτει ομιλήτρια, ε, αυτή, αυτό το αντιφατικό λοιπόν ε, που διαπιστώνουμε δεν μπορεί να εξηγηθεί με λόγους υγειονομικούς. Δηλαδή είναι σαν να ε, κάνει, να ασκεί πολιτική υγεία, υγείας Ευρωπαϊκή Ένωση διαφορετική εντός των συνόρων και εκτός των συνόρων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνουμε με μία μικρή συζήτηση. Σας παρακαλώ, λόγω της περασμένης ώρας, να είστε πάρα πολύ σύντομοι. Η κυρία Γιάλα, πολύ ε, σύντομα κύριε Πρόεδρε και εγώ ευχαριστώ το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεση αυτή, για τις διευκρινήσεις και σίγουρα να πω ότι είμαι, τη συμφωνώ με τις προτάσεις της ε, εισηγήτριας. Πολύ μεγάλη πρόοδος ποιοτική έχει επιτευχθεί σε αυτό το τομέα τα τελευταία χρόνια. Έχουμε προώθηση ε, του ευρωπαϊκού κρασιού στις αναδειόμενες αγορές στο εξωτερικό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά και κατανοώ πλήρως πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια πολιτική συνεκτική, να μην έχουμε επιπρόσθετες φυτεύσεις ε, και τελικά αυτό να λειτουργεί κατά του ανταγωνισμού και κατά της, ε, της ανταγωνιστικότητας δηλαδή, των προϊόντων μας στο εξωτερικό και κατά της ποιότητας των προϊόντων μας. Η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να μας βοηθήσει και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει ε, ως προς τις τοποθετήσεις αυτές. Δηλαδή ότι από τη στιγμή που έχουμε συγκεκριμένη δυνατότητα, ικανότητα σήμερα να εξάγουμε περισσότερο, αναγνωρίζονται τα κρασιά μας περισσότερο στο εξωτερικό, και σε αυτό αναφέρεται και το ελεκτικό συνέδριο στο σημείο 60. Τότε, υπ' αυτή την έννοια, ε, πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβλέψει ε, αυτό κάτι το θετικό. Αυτή τη στιγμή το κάνουμε με την εκβιομηχάνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όχι όμως εδώ, σε αυτό το τομέα και είμαστε σε κρίσιμο σημείο στην κοινή γεωργική πολιτική. Δηλαδή η Ευρώπη αποδεικνύεται πολύ πιο ανταγωνιστική πλέον σε αυτό το τομέα της οικονομίας και τα μέτρα που εφαρμόστηκαν μπόρεσαν να καταστήσουν τον ευρωπαϊκό κλάδο πιο ανταγωνιστικό, τον αμπελοϊνικό δηλαδή, μαζί ε, διατηρώντας παράλληλα τον ποιοτικό χαρακτήρα και ε, αναπτύσσοντας δραστηριότητες marketing. Έχει προβλέψει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα εμπορικό σήμα ποιότητας με το όνομα Ευρώπη για να βγούμε πιο ξεκάθαρα έξω στον κόσμο, όπως το αναφέρει και το σημείο 60 της έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου. Θα πρέπει να υπερπηδήσουμε τις αντιφάσεις, τις εντάσεις εκατέρωθαν και να μπορέσουμε να δρομολογήσουμε αυτό το ευρωπαϊκό σήμα ποιότητας για τα κρασιά ποιότητας πραγματικά και να είναι αυτό εμφανές και στο εξωτερικό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να είμαι σύντομη, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πολύ καλή έκθεση, συμφωνώ. Το καθεστώς εκρίζωσης θέλει να μειώσει τα διαρθρωτικά πλεονέασματα. Όμως, ελοχεύει ο κίνδυνος, ο μόνιμος κίνδυνος εξαφάνισης αμπελώνων, οι οποίοι είναι βιώσιμοι και οι οποίοι είχαν ήδη αναδιαρθρωθεί και μεταρρυθμιστεί. Η πολιτική αναδιάρθρωση των απολώνων είναι πολύ σημαντική για να έχουμε αποτελεσματική αξιοποίηση των ενισχύσεων και της υποστήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ε, δεδομένης της υψηλής ζήτησης για εκρήγηση, δεχομένως μπορούσαμε να έχουμε λιγότερο, με, όχι τόσο μεγάλη ενίσχυση. Έχουμε σαφείς δείκτες, για τις επιδόσεις και πρέπει να τους χρησιμοποιήσουμε. Νομίζω ότι δεν έχουμε βασιστεί σε επαρκή ε, ερευνητικά στοιχεία. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να βοηθήσει τους μη ανταγωνιστικούς αμπελοργούς να εγκαταλείψουν τον τομέα ελοχεύει μεγάλος κίνδυνος να κλείσουν παραδοσιακοί, πολύ σημαντικοί αμπελώνες, οι οποίοι είναι χρήσιμοι όχι μόνο για το κρασί, αλλά και για τη διατήρηση πολιτισμικών στοιχείων εξαιρετικά σημαντικών στην εκάστοτε περιοχή. Και πολύ φοβούμαι ότι στις παραδοσιακές αμπελουργούς χώρας, όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία, τελικά θα μείνουν μόνο οι πολύ μεγάλοι οίκοι, οι πολύ, τα πολύ μεγάλα ε, εινοπία θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των μικρών αμπελουργών και παραγωγών και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι η μικρή εκμετάλλευση, η μικρή γεωργική επιχείρηση είναι αυτή η οποία σέβεται και ακολουθεί πραγματικά τις επιταγές της ποιότητας. Αυτό σίγουρα ισχύει στη Τσεχία, εν πάση περιπτώσει. Είναι πολύ προβληματική η απόφαση να συνεχιστεί η προστασία των δικαιωμάτων φύτευσης και μάλιστα σε τόσο μεγάλο βάθος χρόνου. Θα πρέπει να συζητηθούν όλα αυτά. Ναι, είναι δυνατό να μας βοηθήσει αυτό να ρυθμίσουμε καλύτερα τη γεωργική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την αμπελοϊνική δραστηριότητα. Όμως, σε κάθε περίπτωση, η μικροαμπελουργή και η μικροϊνοπαραγωγή θα πρέπει να βοηθηθούν για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν την βοήθεια της Ευρώπης και στο μέλλον. Χαίρομαι, διότι έχουν υποθεί όλα αυτά, έχουν λεχθεί όλα αυτά και θα πρέπει να υπογραμμίζουμε όχι μόνο τις εξαγωγές του ευρωπαϊκού κρασιού, αλλά να προβλέπουμε και μέτρα στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ενισχύσουμε την κατανάλωσή τους για να βελτιώσουμε την ε, θέση που καταλαμβάνουν στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Τσέσκοβα. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ως προς την παρουσίαση της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου, θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ε, βασική ενδεχομένως διαφωνία. Υπόθηκε ότι το σημείο ανισορροπίας γίνεται όλο και πιο μεγάλο μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ενώ εμείς αυτή τη στιγμή παριστάμεθα ενώπιον ενός προβλήματος στην τροφοδοσία του κρασιού. Πέρσι είχαμε πολύ περιορισμένη σοδιά, μεταξύ άλλων και διότι εξαλείφθηκαν μεγάλες εκτάσεις στην Ευρώπη. Φέτος πάλι θα έχουμε πολύ περιορισμένη εισόδια γιατί ε, πολλές επιφάνειες έχουν επίσης εκριζωθεί τα αμπέλια εκεί. Έχει συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. 150 εκατομμύρια εκατόλιτρα λοιπόν είναι η παραγωγή. Αναμφίβολα φέτος θα χάσουμε αγορές του εξωτερικού διότι δεν θα μπορέσουμε να τις τροφοδοτήσουμε παρκώς με το κρασί που παράγουμε. Και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Ο αμπελοϊνικός τομέας ε, είναι ένας τομέας όπου έχει μειωθεί η κατανάλωση κρασιού στις μεγάλες αμπελοπαραγωγικές και ίνοπαραγωγικές χώρες, κυρίως στην Ισπανία και στην Ιταλία, λιγότερο στη Γαλλία. Αυτό ισχύει. Όμως, η εξάλληψη της απόστασης κρίσης της αγορές επέτρεψε τελικά να πολλαπλασιαστούν οι εξαγωγές. Από 15 εκατομμύρια εκατόλιτρα σε λίγα χρόνια φτάσαμε στην εξαγωγή 23 εκατομμυρίων εκατολίτρων σε τρίτες χώρες. Αυτή είναι μια τάση στην οποία δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε φέτος γιατί δεν υπάρχει κρασί. Δεν υπάρχει αρκετό κρασί. Είπα αυτή την έννοια λοιπόν. στι συζητήσει με το ελεγκτικό συνέδριο έχουμε παρουσιάσει τι αμφιβολίε μα εδώ και αρκετού μήνε για αυτή την ανισορροπία. Τότε αμφιβάλαμε, τώρα είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει αρκετό κρασί. Αυτό τώρα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία χρονιά κατά την οποία ε, να συγκλίνουν κατά τον ίδιο τρόπο διάφοροι παράγοντε, ώστε τελικά να επιτευχθεί πολύ υψηλή απόδοση σε διάφορε χώρε και να αλλάξει και η συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ κατά τον τρόπο των αναλογούντα ώστε να έχουμε εξαγωγές πολύ περισσότερες ή το αντίθετο επίσης να συμβεί, να καταβαραθρωθούν. Αυτά μπορεί να γίνουν. Εν πάση περιπτώσει, η το αντιθετο πίσω να συμβει να καταβαραθρωθουν αυτα μπορει να γινουν εν παση περιπτωσει η ανταγωνιστικοτητα του ευρωπαϊκού κρασιού που ήταν βασικός στόχος της μεταρρύθμισης έχει βελτιωθεί. Και ε, η τα μέτρα της αγοράς ουσιαστικά ε, έκαναν τους, τους συνοπαραγωγούς να αντιδράσουν και να πολλαπλασιάσουν τις εξαγωγές τους. Τώρα λοιπόν θέλω να πω να μπω σε κάτι που έχει επανειλημμένως αναφέρει το ελεκτικό συνέδριο, όπως και η συγγήτρια του Κοινοβουλίου. Εμείς δεν θεωρούμε ότι υπάρχει καμία αντίφαση μεταξύ των δύο βασικών μέτρων της μεταρρύθμισης, δηλαδή μεταξύ της εκρίζωσης, η οποία βοήθησε τους μη ανταγωνιστικούς άμπελοκαλλιεργητές και παραγωγού να βγουν από την αγορά του κρασιού, μεταξύ της εκρίζωσης από τη μία και της αναδιάρθρωσης του αμπελώνα, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει ε, αντίφαση γιατί η αναδιάρθρωση του αμπελώνα επέτρεψε σε συγκεκριμένους συνοπαραγωγούς να γίνουν ανταγωνιστικοί. Στο Languedoc, στη Σικελία, στην Καστήλη Λαμάντσα υπάρχουν ίνοπαραγωγοί που αναδιάρθρωσαν τον αμπελώνα τους και έγιναν ανταγωνιστικοί, έγιναν επαρκείς και πουλάνε το κρασί τους στην αγορά της Ρωσίας, τον είπα ή αλλού και δεν το πάνε το κρασί τους για απόσταξη. Δεν είναι λοιπόν αντιφατικά μεταξύ τους αυτά τα δύο μέτρα η εκρίζωση και η αναδιάρθρωση. Διότι η αναδιάρθρωση μεταξύ άλλων δεν οδήγησε σε τόσο μεγάλη αύξηση της απόδοσης αλλά σε μείωση της απόδοσης μάλιστα και κυρίως αυτό ισχύει στην Ιταλία όπου έχουμε αμπελώνες εξαιρετικά υψηλής απόδοσης και εξαιρετικά κακής ποιότητας. Εκεί έγινε πλήρης αναδιάρθρωση για να βελτιωθεί τα μάλα η ποιότητα και στην Ισπανία. Η μετατροπή δεν αύξησε την απόδοση. Παράλληλα με τη, μετατροπή, με τη ορισμένοι είναι ο παραγωγή με δικά τους λεφτά ε, έκαναν έργα άρδευσης και έτσι στους δικούς τους αμπελώνες βελτίωσαν την παραγωγή τους και μπόρεσαν να εξάγουν σε αγορές του εξωτερικού. Για εμάς το μείγμα των μέτρων ήταν εξαιρετικά θετικό. Θα μπορούσαμε να είχαμε ενισχύσει την εκρίζωση λίγο λιγότερο, είναι το ερώτημα. Ενδεχομένως ναι είναι η απάντηση. Ε, κατά μέσο όρο 10% ε, περισσότερο επιδοτήσαμε και ενισχύσαμε την ε, εκρίζωση συγκριτικά με την προηγούμενη μεταρρύθμιση. Όμως πετύχαμε το στόχο μας πάνω από 170.000 εκτάρια. Από εκεί και πέρα. Λέτε, ή μάλλον να διευκρινίσω και το εξής το μέτρο της εκρίζωσης ήταν ένα προσωρινό μέτρο τα τρία πρώτα χρόνια της μεταρρύθμισης. Δηλαδή, όραμα έχουμε με τη μεταρρύθμιση είναι το όραμά μας είναι να βοηθήσουμε ορισμένους άμπελο παραγωγούς να βγουν από τον τομέα διότι δεν είναι ανταγωνιστικοί και δεν μπορούν να βγουν μόνοι τους και από την άλλη να ενισχύσουμε το κλάδο με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Η εκρίζωση τελείωσε το 2011. Δεν επιδοτείται η εκρίζωση πλέον. Να, κάθε χάσω την Τσέχα βουλευτή. Δεν επιδοτούμε, δεν ενισχύουμε πλέον την εκρίζωση από το 2011 και μετά. Και θέλουμε βέβαια να δουλέψουμε για μια νέα κοινή γεωργική πολιτική. Τώρα, ως προς την προώθηση του κρασιού, θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής. Με δύο διαφορετικούς τρόπους γίνεται αυτό. Η οργάνωση της αγοράς κρασιού επιτρέπει την προώθηση σε τρίτες χώρες του κρασιού και είναι ένα μέτρο με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ήταν ένα νέο μέτρο, το οποίο μάλιστα καθυστέρησαν να εθετήσουν τα κρατη αυτή τη στιγμή όμως το εφαρμόζουν και με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο θα έλεγα. Και ισχύει και ε, σε υφιστάμενες αγορές και σε νέες αγορές. Εξού και οι δείκτες για, την, για τις εξαγωγές των κρασιών είναι εξαιρετικά θετικοί. Έχουν πολύ θετικό πρόσωπο προς το παρόν. Έχουμε όμως μέτρα και για την πρόθεση του κρασιού στις κοινοτικές χώρες. Εξού και στο πρόγραμμα προώθησης των γεωργικών προϊόντων, το οποίο είναι ένα οριζόντιο πρόγραμμα και αναφέρεται και αφορά όλα τα γεωργικά προϊόντα. Κάθε χρόνο έχουμε υποπρογράμματα για το κρασί, τα οποία τονίζουν τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του κρασιού και την ποιότητα των ευρωπαϊκών κρασιών είναι κάπως διαφορετικό από την κοινή οργάνωση κρασιού, γιατί δεν μπορούμε να προωθήσουμε εκεί μάρκες, αλλά την έννοια, το προϊόν κρασί γενικότερα, το προϊόν ευρωπαϊκό κρασί. Έχουμε μέτρα λοιπόν για την προώθηση του κρασιού, του ευρωπαϊκού κρασιού στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Κάθε χρόνο ε, υλοποιούνται τέτοιου είδους προγράμματα. Σχολιάστηκε και το εξής αυξανόμενη επιρροή τρίτων χωρών με τιμές κρασιού εξαιρετικά χαμηλές. Οφείλω να πω το εξής. Δυστυχώς, στον κόσμο, η πιο φτηνή τιμή κρασιού στον κόσμο είναι μια τιμή που αναφέρεται σε ένα κρασί της δικής μου χώρας, ένα ισπανικό κρασί. Δυστυχώς. Πράγματι ισχύει. Υπάρχουν κρασιά φτηνά και είναι φτηνό το κρασί των τρίτων χωρών αλλά όχι τόσο φτηνό όσο η πλειονότητα των ισπανικών κρασιών και κρασιών άλλων χωρών. Άλλωστε έχουμε πολλά ε, κρασιά ευρωπαϊκά που είναι εξαιρετικά φτηνά. Εμάς μας ενδιαφέρει να προωθήσουμε την ποιότητα και θέλουμε να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας λιγότερο στην ποσότητα και περισσότερο στην ποιότητα. Για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό να ανταγωνιστούμε τις τρίτες χώρες που δεν έχουν περιορισμού στα δικαιώματα φύτευσης και που ήδη έχουν το 50% του μεριδίου της αγοράς. Τα ευρωπαϊκά κρασιά σε χώρες πολύ σημαντικές έχουν χάσει σημαντικό μερίδιο αγοράς που είχαν παρά το ότι έχουν αυξηθεί οι εξαγωγές μας. Αυτό ισχύει για τη ΣΥΠΑ, για το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία πολύ λιγότερο, αλλά εν πάση περιπτώσει τα κρασιά μας τα πάνε θαυμάσια, καταπληκτικά, ε, σε αγορές όπως είναι η κινέζικη αγορά. Τελευταίο ερώτημα να το διευκρινίσω. Τα δικαιώματα φύστευσης είναι μια μεταβατική πολιτική. Η μεταρρύθμιση του κρασιού το 1999 έγινε μετά την απόφαση του Συμβουλίου Υπουργών του 1999 και αυτό καταργήθηκε, αποφασίστηκε η κατάργηση το 2010. Με τη σημερινή μεταρρύθμιση αποφασίσαμε να καθυστερήσουμε, να μετακυλήσουμε χρονικά την κατάργηση του συστήματος. Το παρατείναμε. Η απόφαση να τελειώνουμε με τα δικαιώματα εφήτευσης έχει ληφθεί προηγουμένως, στο παρελθόν, όπως σας αναφέρω τώρα. Και αποφασίσαμε απλά να την καθυστερήσουμε για άλλη μια φορά, να την μετακυλήσουμε για λίγο. Ο Επίτροπος κ. Τσιόλος αποφάσισε να συστήσει μια ομάδα υψηλού επίπεδου για το θέμα αυτό τον Μάρτιο. Έχει ήδη συνεδριάσει τρεις φορές η ομάδα υψηλού επίπεδου για τα δικαιώματα φύτευσης και θα καταλήξει στην έκθεσή της η οποία θα παρουσιαστεί ε, στα τέλη του Νοεμβρίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει ως παρατηρητή σε αυτή την ομάδα υψηλού επίπεδου και έτσι ο αντίκτυπο της ενδυνάμει απελευθέρωσης των δικαιωμάτων φύτευσης και στον κλάδο του κρασιού και ε, στους ε, αμπελουργούς. Επομένως θα έχει ο Επίτροπος Τσιόλος την έκθεση, του, την έκθεση αυτή μέσα σε έναν ή δύο μήνες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Να δώσω το λόγο στην εισηγήτρια για να μας κάνει τα δικά της καταληκτικά σχόλια, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές ότι πράγματι η αγορά έχει βελτιωθεί. Δεν πρέπει να είμαστε απεσιόδοξοι και θα πρέπει να, έχουμε, να πάρουμε υπόψη μας και το θέμα της αλλαγής των κλιματικών συνθήκων. Είναι συγκυριακό. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι το κλίμα του χρόνου, του αντίχρονου ε, και ποια επίπτωση θα έχει αυτό στην εκάστοτε σοδιά. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τη γνώμη των ε, κρατών μελών. Και τελικά Δεν ξέρω αν θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητα των παραγωγών και αν θα μειωθεί τελικά και η ποιότητα του κρασιού. Καλό θα είναι να κάνουμε το παν ε, για να, να έχουμε ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αυτά θέλω να πω για να κλείσει το ζήτημα, η συζήτηση του, του ζητήματος αυτού σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Το ελεγκτικό συνέδριο πολύ σύντομα παρακαλώ γιατί το λεωφορείο περιμένει τους συναδέλφους που πρέπει να πάνε στο Λουξεμβούργο. Στην έδρα σας. Ελεγκτικό συνέδριο έχετε το λόγο, αλλά πολύ σύντομα. Μάλιστα, θέμα λοιπόν και εγώ σύντομος. Ε, σύντομες παρατηρήσεις για την γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει κάποια αστάθεια Όμω, όσον αφορά τι καιρικέ συνθήκε, οι καιρικέ συνθήκε ήταν άσχημε τα τελευταία χρόνια και αυτό επηρέασε την παραγωγή κρασιού. Ελπίζουμε να βελτιωθούν οι καιρικέ συνθήκε και ταυτόχρονα να βελτιωθεί και η παραγωγή. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Δεν έχει λυθεί. Αυτό που ζητούμε εμείς από την Επιτροπή είναι μία μακρο, μέσο και μακροπρόθεσμη αξιολόγηση της κατάστασης. Έπειτα η αύξηση της παραγωγής είναι ένα θέμα που μας προβληματίζει ακόμα. Έχουμε τώρα στα σημεία 8 και στα γραφήματα 8 και 9. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι μας μίλησε για τα μέτρα βελτίωσης στα γραφήματα 8 και 9 και εκεί φαίνονται οι επιπτώσεις ξεκάθαρα και στο σημείο 28 οι αναδιαρθρώσεις. Έπειτα να σας ανακοινώσω ότι το, ελεκτικό συνέδριο αυτή τη στιγμή εξετάζει το ζήτημα της ε, διαφήμισης και ελπίζω να έχουμε γρήγορα τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής. Θα σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Τώρα θα ήθελα να κλείσω λοιπόν και το σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης. Αυτή τη στιγμή θα γίνει συνάντηση των συντονιστών, αλλά θα διαρκέσει μόνο δύο λεπτά. Θα ασχοληθούμε αύριο με τα υπόλοιπα ζητήματα. Σας παρακαλώ όσοι δεν χρειάζεται να βρίσκεστε εδώ να φύγετε όσο το δυνατόν συντομότερα και αν ακούνε οι συντονιστές έχουμε μία πρόταση για μία κρόση και για ε, επισκέψεις αντιπροσωπιών. Αυτές οι προτάσεις προετοιμάστηκαν από τις γραμματείες και από το επιτελείο της ομάδας. Το ζήτημα είναι αν συμφωνείτε με αυτές τις προτάσεις. Αν ναι, τότε μπορούμε να τις μεταδώσουμε στις ε, υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.